Um, Καλημέρα συνάδελφοι. Θα ξεκινήσουμε με το σημείο 8 της ημέρας διάταξης παρουσίαση της εκθέσεως του Τζοβάνι Πετρέλη ε, της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας της Ασίας Δεδομένων. Καλώς ήρθες Τζοβάνι που θα παρουσιάσει την ετήσια έκθεση του 2015. Θα έχετε λάβει ηλεκτρονική εκδοχή της εκθέσεως και υπάρχουν και έγγραφα στο χαρτί στην είσοδο το 2015 ήταν ε, πάρα πολύ σημαντικό έτος στην προστασία των δεδομένων για συμφωνίες μεταξύ των διαφόρων φορέων νομοθετήσεως για το πακέτο για προστασία των δεδομένων. Η έκθεση λοιπόν θα καλύψει παραγωγικότατο έτος για το EDPS όσον αφορά εποπτεία και διαβούλευση. Και εσύ Τζοβάνι εδώ να παρουσιάσεις ε, αυτές τις δραστηριότητε. Να σου πω ότι από το διορισμό σου ε, είχε εμφανιστεί στην Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών επανειλημμένα όταν συζητούσαν τα μέλη, το PNR, το TTIP, τη Συμφωνία Αιγίδα και την ακρόαση για την προστασία της ιδιωτικότητας, τη θωράκιση της ιδιωτικότητας. Ε, από ό,τι καταλαβαίνω θα αναφερθεί στη Δευτέρα στο θέμα αυτό για την ασπίδα όσον αφορά την προσωπική ζωή, τα προσωπικά δεδομένα. Είχαμε και αντιπροσωπεία στη Ουάσιγκτον, πήγε την περασμένη εβδομάδα και στο Σαν Φρανσίσκο. Και τα μέλη ε, θα θέλουν να υποβάλουν ερωτήσεις ε, σχετικές. Σε ευχαριστώ που ήρθες, χωρίς να χρονοτριβήσω, σου δίνω το λόγο για ένα δεκάλεπτο, αν συμφωνείς, και μετά θα αρχίσει η συζήτηση. Ευχαριστώ Πρόεδρε, καλημέρα αξιότιμα μέλη της Επιτροπής. Σας ευχαριστώ που για μια ακόμη φορά μου δίνετε δυνατότητα να σας παρουσιάσω την πιο πρόσφατη ετήσια έκθεση ε, της Ευρωπαϊκής Εποπτικής ε, Αρχής για τα προσωπικά δεδομένα. Είναι καινοτόμα περιεκτική έκθεση ε, και αναφέρει τις επιδόσεις, τους δείκτες επιδόσεων και στατιστικά στοιχεία στα παραρτήματα. Ο πολύ καλός συνάδελφος Βοίτσοφ Πεβερόφσκι και εγώ είμαι θα ευγνώμονας όσον αφορά το προσωπικό μας για το αποτέλεσμα. Εδώ και δύο χρόνια περίπου είχε αναφερθεί ότι η γενιά της χιλιετίας ξοδεύει περίπου 18 ώρες την ημέρα καταναλώνοντας ΜΜΕ, ε, στέλνοντας μηνύματα, παίζοντας στο διαδίκτυο, στα κοινωνικά μέσα. Ε, οπότε πρέπει να προφυλάξουμε τη ζωή μας τη διαδικτυακή και είναι κάτι εξίσου σημαντικό αυτό όσο και η προστασία των ανθρώπων στον φυσικό κόσμο και αυτό η Ευρωπαϊκή Ένωση και ο ευρύτερος κόσμος ο, χρωστούν μεγάλο χρέος, έχουν μεγάλη υποχρέωση στο Ευρωκοινοβούλιο, διότι δείξατε ε, πρωτοβουλία, θεσπίσατε φιλόδοξους στόχους για το περιβάλλον το διαδικτυακό. Καταρχάς, από τι φόρο τιμή σε εσάς, ε, Πρόεδρε, στον εισηγητή, στους και και για το GDPR και την οδηγία την προστασία των δεδομένων για την αστυνομία και την ε, ποινική δικαιοσύνη. Πέρσι ήταν το πρώτο πλήρες έτος της θητείας μας. Η λογοδοσία είναι η σημαντικότερη καινοτομία στο GDPR ε, και θα πρέπει να σας λογοδοτεί. Και ο Βόιτσες Μποβορόφσκι και εγώ ε, σε λιγότερες από 100 ημέρες από το διορισμό μας εκπονήσαμε στρατηγική πενταετή. Με αυτή τη στρατηγική στερνιστήκαμε την εντολή που μας αναθέσατε και τη μετατρέψαμε σε πραγματικές δράσεις ε, εκπροσωπεύοντας, ε, εκπροσωπώντας μάλλον στο ύψιστο επίπεδο ε, τη βούλησή σας και δημιουργώντα σχέσει εντό και εκτό τη Ευρωπαϊκή Ενώσεω για αυτόν τον σκοπό. Γι' αυτό εργαστήκαμε σκληρά όλο το έτο για να δημιουργήσουμε συμπράξει και να είμαστε καλοί πρεσβευτέ για τις αξίε και την ελευθερία και τι ελευθερίες της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, κυρίως ενώπιον των ησυχιών και των επικρίσεων. Θέλουμε να είμαστε στην πρώτη γραμμή για τη μεταρρύθμιση και για το δικαίωμα του ατόμου. Ε, είναι ιστορική στιγμή αυτή για την ιδιωτική ζωή και την προστασία των δεδομένων. Σχετικά πρόσφατα η προστασία των δεδομένων ήταν στο περιθώριο για την βιομηχανία της κυβερνήσεις και ίσως και για το κοινοβούλιο τώρα είναι στο επίκεντρο των πολιτικών ζυμώσεων, των δικήσεων, των τεχνολογικών εξελίξεων και η έκθεσή μας προσπαθεί να εξηγήσει ποια είναι η κατάσταση αφορά την προστασία των δεδομένων στην Ευρώπη του 2015. Ε, εξετάσαμε τα θέματα ασφαλής των δεδομένων, τα σύνορα, διοντολογικά θέματα, παγκόσμιες εξελίξεις. Εδώ εξηγούμε πώς εμείς ανεξάρτητος φορέας προστασίας των δεδομένων ε, προσπαθούμε να είμαστε πιο δραστήριοι από ό,τι κατά παρελθόν. Και για να είμαστε ανεξάρτητος φορέας, η προστασία των δεδομένων σημαίνει ότι εποπτεύουμε το πώς γίνεται η επεξεργασία των δεδομένων και δίνουμε συμβουλές στους νομοθέτες πώς θα πρέπει να δρουν για την προστασία των δεδομένων και την προστασία της ιδιωτικής ζωής. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και για τον κανονισμό 45.001 και για τους εθνικούς φορείς της Ευρωπαϊκής Ενώσεως των κρατών μελών. Θέλουμε να έχουμε ψηφιακή προστασία των δεδομένων, διότι αυτό αφορά το πώς επικοινωνούμε, πώς οργάνεται η κοινωνία και πώς λειτουργούν οι επιχειρήσεις, ψηφιακά λειτουργούν. Αφήνουμε, μάλλον ζούμε τη ζωή μας περισσότερο μέσω των διαφόρων συσκευών και των εφαρμογών των διαφόρων ηλεκτρονικών συσκευών και μέσω κινητής εφαρμογής υποβάλαμε σε εσά πέρσι την άποψή μας όσον αφορά τον τελικό γύρο των συνομιλιών για την προστασία των δεδομένων και τη σχετική μεταρρύθμιση. Τώρα το προσωπικό μου με ενημερώνει αξιόπιστα ότι φαίνεται ότι υπάρχουν κάποιες εφαρμογές που μπορούν να αναπτυχθούν, συμπεριλαμβάνουν ε, κάποιες, ε, κάποια κείμενα νομοθετικά για τη διευκόλυνση ε, των αναγνωστών. Είμαστε ο πρώτο θεσμό Ευρωπαϊκή Ενώσεω που διαθέτει σε όλου, βάσει την τσέπη όλων, μια νομική μεταρρύθμιση με παγκοσμίω βελία συνέπεια και μπορείτε να συγκρίνετε δωρεάν τι διάφορε εκδοχέ των κειμένων του GDPR, του GDPR μάλλον, που διαπραγματευόμαστε σε λίγε εβδομάδε. Θα έχουμε επικαιροποιημένη εκδοχή την Τρίτη τη εφαρμογή με την ε, μετά την τελική δοκιμή και θέλουμε να σεβαστούμε το ρόλο των νομοθετών ενώ αναπτύσσουμε παράλληλα και τους πόρους μας ευφυώς και πρακτικώς. Ε, κάποια σχόλια για την ασφάλεια και την ιδιωτική ζωή θα ήθελα να πω ότι στον τόμο 59 της επίσημης εφημερίδας της 4ης ε, Μαΐου έχουμε κάτι που είναι σημαντικό για αυτούς που θέλουν να προστατεύσουν τα θεμελιώδη δικαιώματα και την ιδιωτική ζωή. Πέρασα μια μέρα στην Ευρωπόλ προσφατά για να συζητήσω πώς προετοιμαζόμαστε ούτω ώστε να παίξουμε το ρόλο εποπτικής αρχής και άνοιξε τη διάσκεψη της Europol για την κρυπτογράφηση και την προστασία της ιδιωτικής ζωής όταν ε, αναφέρθηκα, στην έκθεση των συντονιστών στο Συμβούλιο Εσωτερικών και Ασφαλείας ε, για θέματα τρομοκρατίας και είπε ότι δεν υπάρχει σωστή ε, διαβίβαση πληροφοριών μεταξύ των κατανομενών. συζήτηση για το PNR μας υπενθυμίζει ότι πολλά ακόμα θα πρέπει να γίνουν ώστε να βρούμε ειλικρινή ισορροπία μεταξύ των φορέων επιβολής του νόμου και τις δυνατότητες που έχουν στην πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα και από την άλλη πλευρά την προστασία της ιδιωτικής ζωής. Για να το βοηθήσουμε αυτό το θέμα να το προωθήσουμε. Εμείς θα ετοιμάσουμε συμβουλευτικό έγγραφο και ένα σχέδιο εργαλειοθήκη που ανακοίνωσα πέρσι για να βοηθήσουμε τους νομοθέτες ώστε να αξιολογήσουν στην πρακτική την αναγκαιότητα των μέτρων που θα παρεμβαίνουν με τα δικαιώματα όσον αφορά την προστασία των δεδομένων και τη ιδιωτική ζωή. Θα προτείνουμε μια μέθοδο που θα συνοδεύεται από την ομολογία για να εξισορροπηθούν οι διάφορε προτεραιότητε. Και πριν ολοκληρωθεί το έγγραφο αυτό, θέλουμε να ακούσουμε τι απόψει σα και αυτέ τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή και του Συμβουλίου και των εξωτερικών εμπειρογνωμών όσον αφορά την χρησιμότητα των λόγων εγγράφου. Τώρα τι γίνει τη συνεργασία με τους διάφορους φορείς. Εμείς είμαστε ικανοποιημένοι και χαιρόμαστε ότι είδαμε ότι κάποιες συστάσεις όσον αφορά το, την οδηγία του GDPR και την αστυνομία έγιναν δεκτές, όπως η σύστασή μας, δηλαδή να αφήσουμε περιθώριο, ούτω ώστε ανεξάρτητοι φορεί να δίνουν προσανατολισμό όσον αφορά το πώς θα εφαρμόσουμε πρακτικά τα διάφορα προτινόμενα μέτρα. Ο αριθμός των κατοξιδότηση πράξεων ε, μειώθηκε από 48 στην πρόσφατη πρόταση σε 13, ούτως ώστε τώρα έχουμε νέα ζήτηση για διάφορους ε, φορείς αρμοδίους να κινούνται τάχιστα και να είναι αποτελεσματικοί. Και οι αρχές για να συνεργάζονται καλύτερα, οι αρμόδιες, ο, ο κανονισμός έχει δημιουργήσει νέα φορέα, τον EDDB, EDDB, ε, για να διευκολύνει την διαδικασία. Θεωρούμε λοιπόν το GDPR είναι η αφετηρία, ο φορέας μας, δεν είναι κάτι τέλειο, αλλά έχουμε εντοπίσει μαζί με, άλλα, με άλλους συνεταίρους να, τη δυνατότητα να είμαστε έτοιμοι από την πρώτη μέρα με το DPA και θα ετοιμάσουμε και δελτία ε, για τεχνική προετοιμασία ε, που έχει ήδη ξεκινήσει. Είμαστε εδώ σήμερα για να παρουσιάσουμε την ετήσια έκθεσή μας και θέλω να πω ότι είχαμε την καλή τύχη στην αρχή της θητείας μας να κληρονομήσουμε από τους προκατόχους μας ένα γραφείο, μια υπηρεσία που εξακολουθεί να είναι εντάξει, μικρό φορέα αλλά στέρεο και ορίμο. Ε, λοιπόν, θέλουμε να χρησιμοποιούμε σωστά τους πόρους και γι' αυτό υπάρχει ο κατάλληλος έλεγχος όσον αφορά του που μας αντίθεται και έχουμε ζήτηση για συμβουλές όσον αφορά την πολιτική ε, και υπάρχει και ζήτηση και από το δικαστήριο για βασικά θέματα όσον αφορά ε, το δικαίωμα της προστασίας των δεδομένων. Δίνουμε τις συμβουλές και δείξαμε ότι είμαστε ικανοί ε, να δώσουμε τις κατάλληλες συμβουλές και μπορέσουμε να δώσουμε τις κατάλληλες συμβουλές. Έχουμε πολλά στατιστικά στοιχεία τα οποία ίσως μπορούν να παραχθούν και για σας να είναι χρήσιμα να αναφερθώ σε τι στοιχεία των εργασιών μα, ε, σαν φορέα αρμόδιο υποστήριξη των δεδομένων. Καταρχά, κατευθείας γραμμέ για τι κινητέ συσκευέ και ηλεκτρονικέ επικοινωνίε ήταν κάτι που κάλυψε συγκεκριμένε ανάγκε φορέων τη Ευρωπαϊκή Ενώσεω αλλά ήταν αρκετά πρακτικές οι συμβουλές ούτως ώστε να βοηθήσουμε τους ελεκτικούς φορείς. Μετά γνωμοδότηση για τη συμφωνία Ομπρέλα, τη γενική αυτή συμφωνία, θέλαμε να δώσουμε πρακτικές συμβουλές όσον αφορά την βελτίωση της συμφωνίας αυτής και μετά την άποψή μας για το, την πρόταση ε, χρήση πολυφασματικών εικόνων για τη σάρωση των δακτυλικών αποτυπωμάτων ε, για τις ε, ανάγκε του ασύλου. Η οδηγία ε, έχει αφήσει κάποιε ατέλειε Το δικαίωμα της προστασία ιδιωτική ζωής αφορά και την εμπιστευτικότητα των επικοινωνιών και τα τεχνικά μέσα μέσα των οποίων επικοινωνούμε έχουν εξελιχθεί κατά πάρα πολύ μετά την έγκριση της οδηγίας για προστασία της ιδιωτικής ζωής το 2002. Η τρέχουσα αυτή μεταρρύθμιση είναι η άριστη δυνατότητα και ευκαιρία για να προστατεύσουμε περισσότερο την ιδιωτική ζωή και η σημασία δεν είναι ε, οι προσπάθειε δεν είναι διακοσμητικέ, αλλά καταβάλλονται πραγματικέ προσπάθειε για να καλύψουμε τα αγαθά και υπηρεσίε που παρέχονται διαδικτυακά. Θα πρέπει να θέσουμε εν τάξη τον οίκο μα καταρχά. Στο τέλο του έτου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα κάνει κατάλληλε προτάσει για την ε, τροποποίηση του κανονισμού 45-2001. Ήταν παράδειγμα κατά τη ε, θέσπιζε νόμου. Ε, για τα θεσμικά όργανα θα πρέπει να μεταρρυθμιστεί. Μα ζητήσατε να κάνουμε περισσότερα με λιγότερα. Σωστό αυτό λόγω λιτότητας και οικονομικών προβλημάτων. Όραμά μας εξακολουθεί να είναι ένας θεσμός που λογοδοτεί, που καταλαβαίνει τους κανόνες, ε, συμμορφώνεται. Θέλουμε να επικεντρωθούμε επί υποθέσεων που είναι περιπλοκότερες, πιο επικίνδυνες και να δώσουμε τις καλύτερες δυνατές υπηρεσίες στους ανθρώπους. Κλείνοντα, αγαπητέ Πρόεδρε θα ήθελα να πω ότι σα ευχαριστώ, ευχαριστώ όλου σα πάρα πολύ για τη στενή συνεργασία κατά το τελευταίο έτος, ενάμιση έτο, Τίποτα δεν μα δίνει μεγαλύτερη ικανοποίηση σε αυτή τη δουλειά που κάνουμε από το να είμαστε οι πρωταρχικοί σας συνομιλητές, κυρίως όσον αφορά την προστασία των δεδομένων και οι συγκεκριμένα μέτρα. Θα συνεχίσουμε να σας ενημερώνουμε για τη στρατηγική που ακολουθούμε, για τον εξυγχρονισμό την προστασία των δεδομένων στην πράξη, να προωθήσουμε στην πράξη σε παγκόσμιο επίπεδο, να ανοίξουμε ένα νέο κεφάλαιο όσον αφορά την προστασία των δεδομένων. Είμαστε αφοσιωμένοι στην προσπάθεια να βελτιώσουμε την κατάσταση τα επόμενα έτη της θητείας μας για μια ακόμη φορά εκ μέρους των συναδέλφων. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας σήμερα. Σας ευχαριστώ κύριε Μπουταρέλη. Έχουμε δύο εδώ θέματα. τις, ε, τις εκθέσεις ε, για τις εποπτικές δραστηριότητες και τις συμβουλευτικές δραστηριότητες και μια σειρά σημαντικών θεμάτων για τις οποίες γνωμοδοτήσατε. Θα ακούσουμε πρώτα τους συντονιστές. Θα ξεκινήσουμε από την κυρία Χολμάερ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Μπουταρέλη. Περιγράψατε τις διεθνείς δραστηριότητες σας Εμένα θα με ενδιέφερε να μάθω ποιες είναι οι αντιδράσεις των άλλων χωρών έναντι του απόλυτου προτύπου μοντέλου Ευρώπη. Γιατί πολλές φορές άλλες ήπειροι, άλλες χώρες ε, αντιδρούν με έναν τρόπο κάπως ευαίσθητο γιατί θεωρούν ότι ε, εμείς τους δείχνουμε πού θα πρέπει να πάνε, ποια κατεύθυνση θα πρέπει να χαράξουν. Και δεν τους αρέσει αυτό. Οπότε θα ήθελα να μου πείτε πώς είναι οι απόψεις των άλλων, ποιες είναι οι απόψεις των άλλων χώρων. Και ένα δεύτερο θέμα για το οργανωμένο έγκλημα και την τρομοκρατία. Ε, φαίνεται ότι τα επόμενα χρόνια θα υπάρξει μια ε, μεγάλη πρόοδος τεχνολογική, αλγόριθμη ε, τεχνητή νοημοσύνη κτλ. Ποια είναι η γνώμη σας για τον ρόλο της τεχνολογίας τόσο για την προστασία των δεδομένων όσο και για τον εντοπισμό ε, ατόμων που διαπράττουν αδικήματα. Η κυρία Σίπελ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ και για την νέα έκθεση της ε, Υπηρεσίας Προστασίας Δεδομένων. Νομίζω ότι ο μεγάλος αριθμός των δραστηριοτήτων τονίζει για άλλη μια φορά το γεγονός ότι είναι θετικό βεβαίως ότι ε, σε ευρωπαϊκό επίπεδο έχουμε οδηγία και κανονισμό για την προστασία των δεδομένων, αλλά ότι από την άλλη πλευρά βεβαίως δεν έχουν ε, ολοκληρωθεί όλα τα καθήκοντα, όλες οι υποθέσεις. Αντιθέτως, κάθε φορά που ανακύπτει αυτή η συζήτηση, ε, αντιμετωπίζουμε το ζήτημα του κατά πόσο τελικά προστατεύεται η ιδιωτική σφαίρα. Είναι περίπλοκο το θέμα, διότι δεν αρκεί κανείς να αποφασίσει αν σε κάθε επιμέρους μέτρο που έχει ληφθεί εξασφαλίζεται η απαραίτητη ισορροπία. Βεβαίως, ο μεγάλος αριθμός μέτρων ε, έχει ως φυσικό αποτέλεσμα σε έναν βαθμό να περιορίζεται η ιδιωτικότητα. Διάφορα μέτρα λοιπόν, ιδιαίτερα της πολιτικής ασφάλειας, έχουν ε, δημιουργήσει ανησυχίες. Ε, αναφερθήκατε και εσείς στο PNR, στην κρυπτογράφηση, κάτι που μας ενδιαφέρει και μας πολύ. Γνωρίζοντας βεβαίως ότι οι επιτιθέμενοι στο Παρίσι καθόλου δεν αξιοποίησαν κρυπτογράφηση. αντιθέτω, με SMS και κανονικά τηλέφωνα επικοινωνούσαν μεταξύ του. Και βεβαίω η λύση δεν μπορεί να είναι να απαγορευτεί η κρυπτογράφηση. Αντιθέτω, εγώ είμαι υπέρ τη διατήρηση αυτή τη δυνατότητας. Όχι γιατί έχω να κρύψω κάτι, αλλά γιατί θεωρώ ότι η προστασία τη ιδιωτικής σφαίρα και η εμπιστευτικότητα θα πρέπει, είναι κάτι που θα πρέπει να προστατεύεται και στην ψηφιακή σφαίρα. Χθε στην Επιτροπή ε, είχα την ευκαιρία να μιλήσω με τον κύριο Ναβαρέτ από τη Europol και το Κέντρο Καταπολέμησης Τρομοκρατίας και είχα την εντύπωση, είχα μάλλον την ευκαιρία να συζητήσω μαζί του ποιες άλλες δυνατότητες υπάρχουν προκειμένου να μην θέσουμε στο στόχαστρο την κρυπτογράφηση. Τέλος, να σας θέσω και ένα ερώτημα. Έχουμε τώρα τον γενικό κανονισμό και την οδηγία για την προστασία των δεδομένων. Παρόλα αυτά, η Κομισιόν βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις για ε, την αναθεώρηση του, του, του, της ασπίδας ιδιωτικότητας. Μπορείτε να μας πείτε σε τι ακριβώς χρειάζεται αυτό το privacy shield, αυτή η ασπίδα ιδιωτικότητας, παρά το γεγονός δηλαδή ότι έχουμε πλέον ένα γενικό κανονισμό για την προστασία των δεδομένων. Και με ενδιαφέρει ε, αν και πότε εσείς ως ε, Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων πρόκειται να γνωμοδοτήσετε για αυτήν την ε, πρόθεση ή την πρόταση που θα υποβάλει η Κομισιόν. Νομίζω ότι είναι απαραίτητο να υπάρξει και μια δική σας γνωμοδότηση επί των ε, θεμάτων αυτών. Μα μας είπε ότι την Δευτέρα θα γνωμοδοτήσει για το θέμα της ιδιωτικότητας. Κύριε κυρία Έρνστ. Ευχαριστώ και από τη δική μου πλευρά. Σας ευχαριστώ πολύ για το έργο σας. η ψύχρεμη και επικοδομητική συνεργασία που έχουμε όλα αυτά τα χρόνια με τον EDPS είναι πολύ σημαντική για μας. Και ξέρετε ότι είστε πιο απαραίτητος από ποτέ. Δύο θέματα. Έχουμε τον γενικό κανονισμό και την οδηγία που πλέον υλοποιούνται. Βεβαίω αυτό θα διαρκέσει πολλά χρόνια έως ότου ολοκληρωθεί η διαδικασία αυτή στα κράτη-μέλη. Υπάρχουν μέσα ελέγχου, έχετε εσείς τρόπο να εξετάσετε σε ποιο βαθμό και κατά πόσο τα κράτη-μέλη και οι αρχές των κρατών μελών εφαρμόζουν όλα αυτά που προβλέπουν τα δύο, οι δύο αυτές νομοθετικές πράξεις. Το δεύτερο, αποκτήσατε μεγαλύτερες αρμοδιότητες και με τη Europol. Ε, αν τελικά αυτό συνέβη δεν το ξέρω γιατί εμείς είχαμε εκφράσει ε, τις ανησυχίες μας και τις αμφιβολίες μας για το κατά πόσο κάτι τέτοιο θα ήταν εφικτό στην πράξη. Ε, εσείς θεωρείτε ότι έχετε επαρκή στελέχωση, επαρκή πόρους για να ανταποκριθείτε στις αρμοδιότητες που όπως είπα είναι πολύ μεγαλύτερες πλέον. Οι δικές σας. Και τρίτον. Για να είμαστε ειλικρινείς, είναι ε, σαν να ζούμε σε μια πολύ περίεργη ε, ήπειρο, ε, γιατί α, αφενός θεσπίζουμε και αποφασίζουμε για τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Δεδομένων και 30 δευτερόλεπτα αργότερα θεσπίζεται το PNR. Υπάρχει μεγάλο πρόβλημα και μεγάλη αντίφαση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και ε, για την συμφωνία ομπρέλα με τις ΗΠΑ, όπου δεν προβλέπεται τίποτα για τους ανθρώπους που δεν είναι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ποια είναι η γνώμη σας για αυτό το θέμα. Γιατί έχουμε τεράστια προβλήματα. Και νομίζω ότι θα πρέπει να συνεχιστεί η συζήτηση για, τα αυτά, για αυτά τα θέματα. Ε, συνεδριάζουμε και με τους ε, συντονιστές, με τους σκιώδεις, για ε, το ζήτημα αυτού του, αυτής της συμφωνίας ομπρέλα και θα ήθελα να μου πείτε ε, ε, πολύ ειδικά τη γνώμη σας για τους μη πολίτες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστώ κύριος Μπόνι. Σας ευχαριστώ. Και σας ευχαριστώ για την παρουσίαση κύριε Πόπτη. Θα σας παρουσιάσω τη γνώμη για την έκθεση αργότερα αφού τη διαβάσω πρώτα γιατί δυστυχώς μέχρι τώρα δεν είχα το χρόνο να την μελετήσω πισταμένος. Ο ρόλος ε, του Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας Δεδομένων ε, αυξάνεται. Έχουμε νέες προκλήσεις. στην εφαρμογή της οδηγίας για το PNR, το Μητρό Ονομάτων Επιβατών. Επεξεργαζόμαστε τη νέα οδηγία κατά της τρομοκρατίας. Έχουμε τη συζήτηση για την κρυπτογράφηση με προτάσεις που έγιναν την περασμένη εβδομάδα από την Ευρωπόλ και την Ενίσα. Ε, όλες αυτές οι λύσεις διαμορφώνουν ε, τις ε, απαιτήσεις και τα κριτήρια της νέας ισορροπίας που θα πρέπει να βρούμε μεταξύ της εσωτερικής ασφάλειας και της προστασίας της ιδιωτικότητας. Επίσης, θα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε τα προβλήματα και της ασφάλειας και της ιδιωτικότητας. Έχω μερικές ερωτήσεις. Ποιος είναι ο ρόλος και η ανάμειξη του, του Ευρωπαίου Επόπτη στην εφαρμογή του αυτού του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία των Δεδομένων, του GDPR. Βέβαια δεν είναι τέλειος ο κανονισμός, αλλά πώς θα βρούμε δυνατότητες για πιο ελαστικούς όρους για την επεξεργασία των δεδομένων με κατάλληλες ε, προϋποθέσεις προκειμένου να βοηθήσουμε την επιστημονική πρόοδο και πώς ε, θα καταστήσουμε την εφαρμογή μια λύση που δεν θα καταστρέψει την εναρμόνιση των κανονισμών ε, για την προστασία δεδομένων. Γιατί έχουμε 54 ε, διαφορετικές επιλογές σε εθνικό επίπεδο. Πώς θα έχουμε ένα πιο περιεκτικό και πιο εναρμονισμένο πλαίσιο. Ε, επεξεργάζεται κάποιες κατευθυντήρες γραμμές αυτή τη στιγμή και αν ναι, για ποιους τομείς. Σε ό,τι αφορά τη συζήτηση για την κρυπτογράφηση, πώς την κρίνεται γιατί ανακύπτει η ανάγκη ανέβρεση λύσεων και στον τομέα αυτό. Έχουν κατατεθεί ήδη προτάσει, όπω σα είπα, στην επιστολή τη Ευρωπόλ. Πιστεύετε ότι θα πρέπει να επιταχύνουμε τι εργασίε για την αναθεώρηση τη οδηγία για την ιδιωτική σφαίρα στι ε, ηλεκτρονικέ επικοινωνίε. Και τι, ποια είναι η γνώμη σα για την ασπίδα τη ιδιωτικότητα το Privacy Shield, όπω ρώτησε και κάποια προλαλήσασα ε? Είμαστε στη φάση της διεκπαιρέωσης. Ε, τι μέλη να κάνουμε σε αυτή τη φάση κατά τη γνώμη σας. Δεν ζήτησε άλλος κανείς το λόγο. Η Μαρία... Η Μαρία δεν ξέρω, θέλει άλλος κανείς, όχι. λυπάμαι που καθυστέρησα κάπως, αλλά η πτήση μου με καθυστέρησε. Όπως και άλλοι που με τον κανονισμό, και εγώ διαρωτώ με για τις εξελίξεις και με προβληματίζει ιδιαίτερα το θέμα της συνεργασίας με τις αρχές προστασίας δεδομένων των κρατών μελών. Ποιος είναι ο ρυθμός εφαρμογής αυτού του κανονισμού. Υπάρχουν προβλήματα στην εφαρμογή, υπάρχουν προσκόμματα. Πιστεύετε ότι θα πρέπει εμείς να κάνουμε κάτι περισσότερο τι σα επισημαίνουν οι αρχέ προστασία δεδομένων, Γιατί μια διετία είναι πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, γιατί είναι και περίπλοκο ο κανονισμό. Το ίδιο ισχύει για την οδηγία. Θα χρειαστεί περισσότερο. Γιατί έχει προταθεί και τι ε, αστυνομικέ δυνάμει των κρατών μελών να αντιμετωπίζουν διαφορετικά την προστασία των δεδομένων, να την ενσωματώσουν στα συστήματά του. και δεν είναι όλοι ικανοποιημένοι με αυτή την πρόταση. Ποια είναι η εντύπωση που αποκομίσατε και ποια είναι η εμπειρία σας από την ε, επαφή και την επικοινωνία με τις αρχές και τους φορείς προστασίας δεδομένων στα κράτη-μέλη. Πώς πηγαίνουν τα πράγματα. Ευχαριστώ η Σοφία Έντβελτ. Ευχαριστώ. Δίστασα να ζητήσω το λόγο, γιατί και εγώ έφτασα κάπως καθυστερημένα και ίσως ε, καλύψατε τις ερωτήσεις που θα κάνω ε, να με συμπαθάτε αν έγινε κάτι τέτοιο. Σε ό,τι αφορά την ασπίδα της ιδιωτικότητα, θεωρεί ο Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων ότι η ασπίδα ιδιωτικότητας ε, είναι θωρακισμένη από παραβιάσεις, ατασταλίες. Έχουν γίνει κάποιες μελέτες για να αποφευθούν οι καταχρήσεις και οι εθνικέ αρχέ προστασία δεδομένων ε, μήπω θα, την εφαρμόσουν με διαφορετικό τρόπο, υπάρχουν τέτοιε ανησυχίε. Μήπω κάποιε αρχέ προστασία δεδομένων θα επιτρέψουν τη μεταφορά δεδομένων και άλλε όχι. Γιατί αυτό θα ήταν ε, ε, το απευκταίο, να υπάρχει διαφορετική εφαρμογή αυτή τη ασπίδα τη ιδιωτικότητα. Το δεύτερο θέμα και το αποσύρω το έχετε ήδη καλύψει. Το θέμα του ελέγχου της αναγκαιότητας και της αναλογικότητας. Ξέρω ότι είστε ιδιαίτερα ευαίσθητος για τα θέματα αυτά και θα ήθελα να μου εκφράσετε τα συμπεράσματά σας. Δεν ξέρω τι μπορείτε να μας πείτε για την ασπίδα ιδιωτικότητα. Γιατί τη Δευτέρα θα γίνει επίσημη ανακοίνωση για το θέμα αυτό. Πάντως θα μπορούσατε ίσως κάποια γενικά σχόλια και γενικές αρχές να μας ε, εκθέσετε. Γιατί επίσημα θα γίνει αναγγελία τη Δευτέρα. Τζοβάνι, παρακαλώ, έχεις το λόγο. Ευχαριστώ και ευχαριστώ και τους ευρωβουλευτές ε, για τις ενδιαφέρουσες ερωτήσεις τους. Κυρία Χολμάιρ, όλο και περισσότερες χώρες ασχολούνται με το θέμα της προστασίας των δεδομένων στον κόσμο και από άποψη ψηφιακή εμείς είμαστε ψηφια. Ε, είχαμε 109 χώρες στον κόσμο που εστενίζονται τους νέους κανόνες, τους κανόνες νέας γενιάς ψηφιακούς για την επεξεργασία των δεδομένων. Εμείς ε, ενδιαφερόμαστε περισσότερο για το ευρωπαϊκό μοντέλο από ότι για προηγούμενες προσπάθειες αυτορύθμισης κυρίως. Και πιστεύουμε ότι εξαιτία τη παγκοσμιοποιημένη τάση που υπάρχει, ο τομέας που καθορίζει τη συζήτηση είναι αυτός, ο ψηφιακός. Και ο Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων δεν είναι ιδεώδης ούτε ήταν το όνειρό μου να λάβει αυτή τη μορφή. Πάντως θα τον ε, υπερασπίσω ε, περήφανα και πιστεύω ότι κατ' ουσία είναι σωστός και θα φροντίσω και θα προωθήσω την εφαρμογή του. Γνωρίζω ότι το θέμα βρίσκεται στο επίκεντρο της προσοχής και εκτός της Ευρωπαϊκής ε, Ένωσης. Μερικές φορές προκαλεί έκπληξη, ακόμη και εκνευρισμό, γιατί μερικοί έχουν την αίσθηση ότι εμείς ε, επιβάλλουμε τις αρχές μας ε, για εξοδοφικότητα και ότι προσπαθούμε να εφαρμόσουμε ε, τις δικές μας αρχές ε, σε όλους, άσχετα από το που βρίσκονται οι σερβερ. Αλλά εγώ πιστεύω ότι εμείς πραγματικά πρωτοστατούμε στην συζήτηση που γίνεται διεθνώς και πιστεύω ότι έχει νόημα να περιορίσουμε τη γραφειοκρατία, να επικεντρωθούμε σε ασφαλιστικέ δικλείδε αποτελεσματικέ και όχι σε κριτήρια και απαιτήσει, να αναλύσουμε πώ θα μπορέσουμε να εφαρμόσουμε επιτυχώ αυτού του ρόλου και στον κόσμο των μεγάλων δεδομένων, των big data. Και οι γνωμοδοτήσει μα για τη διοντολογία και για τη συμφωνία πλαίσιο και για τη διαλειτουργικότητα έχουν ήδη δοθεί. Και θέλουμε να εξηγήσουμε ότι ο γενικό αυτό κανονισμό για την προστασία δεδομένων δεν είναι κάτι που μπορεί κανεί να αυτοσχεδιάσει σε λίγε εβδομάδε. Είναι κάτι που σταδιακά θα αλλάξει, αλλά πρέπει να αρχίσουμε να τον εφαρμόζουμε αμέσω. Και τον Ιούλιο θα πάω στη Σιγκαπούρη, Σιγκαπούρη για το φόρουμ ε, του δικτύου των ε, ρυθμιστικών αρχών για την ιδιωτικότητα για να εξετάσουμε την. Ε, ε, σχέση του Γενικού Κανονισμού με άλλες περιφερειακές προσεγγίσεις ε, και να εξετάσουμε κάποιους, ε, και κάποια άλλα εργαλεία όπως είναι οι δεσμευτικοί κανόνες για τις επιχειρήσεις. Και μάλιστα όπως και ο πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών για την ιδιωτικότητα και εγώ προσπαθώ να είμαι πολύ δεκτικός στη συζήτηση και θα πρέπει να δούμε αυτό το θέμα της ιδιωτικότητας ε, και επειδή ακριβώς έχω ε, εμπειρία σε θέματα πάταξης του οργανωμένου εγκλήματος και της μαφίας, θεωρώ ότι οι, οι δικαστικές αρχές θα πρέπει να έχουν πρόσβαση σε διαθέσιμες πληροφορίες, σε νομότυπα φυσικά, με διαφανή τρόπο, ε, με αμοιβέ εμπιστοσύνη και να εφαρμόσουμε με σύγχρονο τρόπο τις αρχές της αναγκαιότητας και της αναλογικότητας. Του τέστην θα πρέπει να υπάρχει μεγαλύτερη σύγκληση προς τις νέες τεχνολογίες και επίσης να αντιληφθούμε ότι η θέσπιση μια νέας βάση δεδομένων δεν είναι από μόνη της ε, η λύση. Γιατί σε μερικές περιπτώσεις η πληθώρα δεδομένων ε, είναι αντιπαραγωγική. Μερικέ φορέ μα λείπει η ανάλυση και δεν μπορούμε να εχωρού, στη λύση των αλγορίθμων την, τον εντοπισμό των εγκληματιών. Μερικές φορές απαιτείται και η ανθρώπινη παρέμβαση, η ανταλλαγή πληροφοριών και μερικές φορές χρειάζεται και εναρμόνιση διαφορετικών λογισμικών και διαφορετικών προσεγγίσεων. Κυρία Ζίπελ, έχετε δίκιο. Έχουμε πολλά μέτρα για την προστασία των δεδομένων και αυτό είναι το αποτέλεσμα μιας ε, οριζόντιας προσέγγισης της προστασίας των δεδομένων. Το ένα θέμα αφορά την κρυπτογράφηση. Εδώ δεν πιστεύω ότι υπάρχει αντιπαράθεση μεταξύ ασφάλειας ε, και ιδιωτικότητας, αλλά είναι θέμα ε, ασφάλειας περισσότερο. Και η κρυπτογράφηση σήμερα είναι αναπόφευκτη από τεχνική άποψη. Δεν υπάρχει εναλλακτική λύση για να προσπίσουμε καλύτερα και να θωρακίσουμε τα δίκτυα και τις πληροφορίες και τις βάσεις δεδομένων μας. Και μάλιστα στην περίπτωση ε, μια υπόθεση ε, του FBI είπα ότι φυσικά θα πρέπει να έχει δικαίωμα το FBI να έχει πρόσβαση σε δεδομένα. Το θέμα είναι ότι δεν μπορεί το FBI να ζητά από μια επιχείρηση να αλλάξει το επιχειρηματικό της μοντέλο, το επιχειρησιακό της μοντέλο και να επιτρέπει σε ολοκληρωτικές κυβερνήσεις ή hackers να έχουν εύκολη πρόσβαση στις συσκευές. Αυτό θα ήταν το τέλος της ασφάλειας στο χώρο εργασίας. Αυτό είχα αποφαθεί και στην περίπτωση FBI κατά της ε, Apple. Τώρα, σε ό,τι αφορά την ΕΝΙΣΑ και το, την Ευρωπόλ, είναι θέμα επιβολής νόμου περισσότερο αλλά κάποια συνετά σχόλια για την κρυπτογράφηση και κάποιες δημιουργικές ιδέες υπάρχουν. Και με τον Rob Wainwright συμφωνούμε με τον διευθυντή της Ευρωπόλ για την ανάγκη να συνεχιστεί η συζήτηση που θα πρέπει να είναι πιο ευρεία. Να μην περιορίζεται μόνο στις συσκευέ και σε διάφορα άλλα εργαλεία, αλλά να δούμε ποιες θα είναι οι συνέπειες και οι βραχυπρόθεσμες και οι μακροπρόθεσμες. Πάντως, βράχει πρόθεσμα, η ασφάλεια δεν θα είναι μόνο αναπόφευκτη, αλλά και νόμιμη υποχρέωση. Και με βάση το γενικό κανονισμό θα πρέπει να υιοθετούνται τα καλύτερα διαθέσιμα μέτρα ασφάλειας. Σε ό,τι αφορά την ασπίδα της ιδιωτικότητα, θα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι οι μεγάλε εταιρείε προσανατολίζονται προ κάποιε στερεότυπε ε, ρήτρε δεσμευτικέ και δεσμευτικέ κανόνε και Λιγότερο από 400 ε, μικρομεσαίες επιχειρήσεις ενδιαφέρονται για μεταφορά δεδομένων σε στρατηγικούς εταίρους όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες. Και όπως είπα, στις 30 Μαΐου θα υιοθετήσουμε σχετική γνωμοδότηση και υπάρχει και μια ειδική ομάδα εργασίας για το θέμα αυτό. Πάντως ε, είναι εύλογες αυτές οι, οι απορίες και οι ανησυχίες. Ε, περιμένουμε τις απαντήσεις και στο μεταξύ πραγματοποίησαμε μία ανάλυση, κυρία Ιντβέλτ, γιατί οι παράμετροι της λύσης δεν είναι μόνο η οδηγία 9546 ε, και η οδηγία πλαίσιο που θα ισχύει μέχρι τις 24 Μαΐου 2018, ε, πρέπει να τις ε, επανερμηνεύσουμε με βάση την υπόθεση ΣΡΕΜΣ και τι σημαίνει ουσιώδες ισοδύναμο και πώς θα πρέπει να γίνει, πρέπει να γίνει έλεγχος του ουσιώδους ισοδυνάμου. Θα πρέπει να σεβαστούμε την ουσία κάθε όρου και απέτηση. Πάντως, η, η δική μας ομάδα εργασίας ε, έκανε αυτή την ανάλυση που θα ολοκληρωθεί εντός ολίγου και θα επικεντρωθούμε σε συγκεκριμένα θέματα όπως είναι η αυτόματη επεξεργασία, το ανεξάρτητο καθεστώς του διαμεσολαβητή, μέτρα αποκατάστασης και μεταφορά. Αυτά είναι μερικά από τα σημεία που εξετάζουμε και θα υιοθετήσουμε δραστήρια και προορατική προσέγγιση παρόμοια με αυτή που υιοθετήσαμε μαζί ε, και για την συμφωνία πλαίσια την Umbrella Agreement. Γιατί η ασπίδα ιδιωτικότητας απαιτεί σημαντικές βελτιώσεις. Και ο ρόλος μας θα είναι δραστήριος και όχι απλώς διακοσμητικός. Θα πρέπει να αναζητήσουμε τις κατάλληλες λύσεις. Κυρία Ένστ, σας ευχαριστώ για τα σχόλια και νομίζω ότι ο κίνδυνος εδώ είναι τι μπορούν τώρα να κάνουν τα κράτη-μέλη. Έχουμε στη γνωμοδότησή μας πέντε κατηγορίες εθνικών διατάξεων σε εθνικό επίπεδο που είναι έμεσες. Ε, αναφέρονται μέσω ε, είτε γίνονται ανεκτές από τον Γενικό Κανονισμό, είτε απαιτούνται από τον Γενικό Κανονισμό. Έχουμε και διατάξεις που δεν αφορούν τη διαδικασία των δεδομένων και το μίσ όπω η επιστημονική έρευνα που αφήνουμε μεγαλύτερη διακριτική ευχαίρεια στα κράτη-μέλη. Εμεί ε, χαρακτηριζόμαστε από επαγγελματισμό. Δεν μα ε, ενδιαφέρει αποπτία σε εθνικό επίπεδο, δεν είναι αυτή η αρμοδιότητα μας. Πάντως εθαρρύνουμε τα κράτη-μέλη να ε, είναι ακριβή και ο Γενικό κανονισμός θα είναι άμεση εφαρμογή. Τώρα σε ό,τι αφορά την λεπτομεριακή εφαρμογή, αυτό αφορά τα κράτη-μέλη. Για την Ευρωπόλ. Σας είμαστε ευγνώμονες για την εμπιστοσύνη και δεν ολοκληρώνεται εδώ διαδικασία γιατί στις αρχές του, νέου, ε, του επόμενου έτους θα υιοθετηθεί ένας νέος κανονισμός και εμείς ενθαρρύνουμε την νομοθετική αρχή να εναρμονίσει το μοντέλο ε, για τους πρώην τομείς του τρίτου πυλώνα και το σύστημα προστασίας δεδομένων. Δεν θα έχουμε απλώς συνεργασία JSA-JSB. Θα πρέπει να έχουμε μία reductio unitatem, Ήρθε αυτή η ώρα. Επίσης δεν έχουμε αρκετούς πόρους και ελπίζω να γίνει δεκτός ο, ο προϋπολογισμός για το 2017, αλλά μπορεί να μην έχουμε πόρους, αλλά ε, γνώσεις έχουμε και έχουμε συνεργασία με το JSB της Ευρωπόλ για να έχουμε αποτελεσματική συνεργασία και ελέγχους. Συμφωνώ για τα σχόλιά σας, αλλά υπάρχουν λύσεις ε, στη Συμφωνία Πλαίσιο για να βρούμε συγκεκριμένες λύσεις. Και μάλιστα και τα μέτρα αποκατάστασης περιλαμβάνονται στη Συμφωνία Πλαίσιο. Και μάλιστα προηγήθηκαν της ε, υιοθέτηση της ε, ε, νομοθετικής πράξης για, δικαστικά, για τα δικαστικά ένδικα μέσα. Δεν είναι απόλυτα ικανοποιητική η λύση, αλλά θα σας εξηγήσουμε στη γνωμοδότηση γιατί δεν μας ικανοποιεί πλήρως. Παρόλο που αυτό δεν έχει άμεση σχέση με το θέμα της ασπίδας Κύριε Μπονή, θα καταφέρετε να διαβάσετε γρήγορα την έκθεση, τη φετινή. 68 σελίδε είναι. Τι κάνει ο Ευρωπαϊο Επόπτη Προστασία Δεδομένων. Εργαζόμαστε 24 ώρε το 24ωρο. Ο Γενικό Κανονισμό αποτελεί μια μεγάλη ευκαιρία και ε, εμείς παρεμβαίνουμε και στην επιστημονική έρευνα. Έχουμε ε, θεσπίσει και ορισμένες συστάσεις για την ομοθεσία που έχουν περάσει οι συνομοθέτες πρέπει να επαγρυπνούμε για το τι κάνουν τα κράτη-μέλη, πότε υπάρχουν παρανοήσεις ή παρεξηγήσεις σχετικά με την προστασία των δεδομένων και πότε κάτι τέτοιο μπορεί να αποβεί ε, εις βάρος της ε, δημόσιας έρευνας. Απάντησα για την κρυπτογράφηση και για την ασπίδα ιδιωτικότητας. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι ελπίζω πραγματικά ότι το άρθρο 30, η Επιτροπή του άρθρου 31 θα καταφέρει να υιοθετήσει γνωμοδότηση για αυτό το θέμα. Ξέρουμε ότι η διαδικασία αυτή βρίσκεται σε εξέλιξη, υπάρχουν κάποιοι συγκεκριμένοι κανόνες επιτροπολογίας, αλλά ελπίζω ε, ε, ότι θα καταφέρει η Επιτροπή αυτή να καταλήξει σε γνωμοδότηση. Επίσης, ε, οργανώνουμε δημόσια διαβούλευση για την, για την ηλεκτρονική ιδιωτικότητα και το άρθρο 35 είναι το άρθρο εκείνο που προστατεύει τις επικοινωνίες στο, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρέπει να διατηρηθεί. Ενθαρρύνω λοιπόν να επικεντρωθούμε στα σημαντικά ζητήματα σχετικά με την ε, τεχνολογία ε, σε ε, ευέλικτα μέσα για να μην προχωρήσουμε σε υπερβολές αλλά είναι σημαντικό να διατηρηθεί αυτή, αυτό το άρθρο 35. Γιατί την κυρία Λόριστη, νομίζω ότι μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι ο γενικός κανονισμός θα στεφτεί με επιτυχία ως προς την ολοποίησή του. Εμείς ε, συνεργαζόμαστε με τις Εθνικές Αρχές Προστασίας Δεδομένων. Στις 10 η ώρα σήμερα θα κάνουμε και μια ε, συνάντηση με τις αρχές αυτές. Ε, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων έχει ως στόχο του να δημιουργήσει πλατφόρμες για τη διμερή και την πολυμερή συνεργασία. Ε, νομίζω ωστόσο ότι το μεγάλο ζήτημα είναι η λογοδεσία. Θα πρέπει όλοι οι φορείς, όλοι οι εμπλεκόμενοι φορεί να ε, ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους. Οι αρχές προστασίας δεδομένων έχουν μεγάλη ευθύνη σε αυτόν τον τομέα. Η λογοδοσία σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωση είναι τεράστιο ζήτημα. εγώ θα συναντηθώ με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, με το Ελεκτικό Συνέδριο, με, ε, με διάφορους φόρους και θα τους καλέσω να αναλάβουν τα ενία σε αυτόν τον τομέα. Γιατί τους αφορά και εκείνου. Και τέλο ερώτηση για την αναγκαιότητα και την αναλογικότητα, κυρία Ίντβελτ εξήγησα στις, στις εισαγωγικές μου παρατηρήσεις ότι σε πολύ λίγες μέρες θα δημοσιεύσουμε το πρώτο έγγραφο σχετικά με αυτό το ζήτημα για την, ε, για το, για την εργαλειοθήκη αναναγκαιότητας και στη συνέχεια θα ε, ε, εκδώσουμε και ένα σχετικό έγγραφο για την αναλογικότητα. Ευχαριστώ λέει ο Πρόεδρος. Να πω επίσης ότι στην ε, αποστολή ε, είχαμε ε, την προηγούμενη εβδομάδα σημαντικότατες συζητήσεις για την ασπίδα ιδιωτικότητας και όλο το πολιτικό φάσμα στις ΕΠΑ παρακολουθεί με μεγάλο ενδιαφέρον ποιο, ποια είναι η άποψη που θα διαμορφώσουμε εμείς εδώ στο Κοινοβούλιο. Οπότε περιμένουμε τη Δευτέρα την έκθεση για το Privacy Shield. Σας ευχαριστώ για το έργο σας στο παρελθόν και στο παρόν και θα ε, συζητήσουμε βεβαίως το ζήτημα αυτό και με αφορμή την έκθεση της ε, αποστολής. Λοιπόν, να προχωρήσουμε στα, στο, στο 9 και στο 10 για τα ευφυή σύνορα. Το Φεβρουάριο του 2013 από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τα σύνορα μετά ανακοίνωση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή το Φεβρουαρίου του 2008 που πρότεινε ότι πρέπει να δημιουργηθεί ένα σύστημα εισόδου-εξόδου ε, στο πρόγραμμα καταχωρήσεως των αξιδιωτών για να κάνω μια ταχεία παρουσίαση πριν παρουσιάσω τον κύριο Δίας Δεμέρα που θα πάρει τον λόγο. Στην πρώτη εξέταση του πακέτου για τα φύση νερό, το Συμβούλιο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέφρασαν διάφορα προβλήματα και ανησυχίε τεχνική φύσεω και δαπανών κλπ. Και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έκανε ένα εγχείρημα ελέγχου του όλου εγχειρήματο σε δύο φάσει. Πρώτα απ' όλα έγινε τεχνική μελέτη, μελέτη του κόστου που ολοκληρώθηκε τον Οκτώβριο του 2014 και δεύτερον έγινε μια φάση 12 μήνη δοκιμών που ανέθεσε στο Ελίσσα η Ευρωπαϊκή Ένωση και ολοκληρώθηκε τον Νοέμβριο του 2015. 6 Απριλίου του 2016 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέτησε αναθεωρημένη νομοθετική πρόταση που αποτελείται από κανονισμό για τη δημιουργία ενός συστήματος εισόδου-εξόδου και πρόταση τροπολογίας του κώδικα συνόρων Σέγγεν για να γίνουν εναγκαίες τεχνικές αλλαγές, ούτως ώστε να δημιουργηθεί το σύστημα εισόδου-εξόδου. Έκανα αυτή την παρουσίαση για να επικαιροποιήσω τις γνώσεις εκείνων που θέλουν να ασχοληθούν το περίπλοκο θέμα. Έχουμε εδώ τον Δίας Δεμέρε, τον εισηγητή μας και θέλω να του δώσω το λόγο πρώτος να μιλήσει εκείνος πριν γίνει η παρουσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, εκτός αν θέλετε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μιλήσει πρώτη. Τι θέλετε να κάνετε, πρώτος εσείς, πρώτη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Προτιμώ να μιλήσει πρώτη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, κύριε Πρόεδρε. Okay, so we... Καλώς. Στρεφόμαστε προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, λοιπόν, για να προβεί στην παρουσίασή της. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ο κ. Ρόζενμπεργκ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Το πακέτο του 2016 φύση Σύνορα υιοθετήθηκε σε 6 Απριλίου. Εμπεριέχει τρία στοιχεία. Πέρα από την πρόταση για τη δημιουργία συστήματος εισόδου-εξόδου και τις αναθεωρημένες προτάσεις για τροποποίηση του κώδικα συνόρων του Σέγγεν είχαμε και ανακοίνωση για ισχυρότερα και φέστερα συστήματα πληροφοριών για την ασφάλεια των συνόρων και ανακοίνωση παρουσιάστηκε σε πρώτη συνεδριασή σας, δεν θα αναφερθώ σε αυτό τώρα. Θέλω να πω ότι αποτελεί ένα κομμάτι του πακέτου. Πριν υπησέλθω σε λεπτομέρειε να επενθυμίσω κάτι σύντομα, να αναφερθώ στην φάση προετοιμασία ήδη, είπατε ότι το όλο θέμα έχει μακρά ιστορία και αναφερθήκατε και στο όλο εγχείρημα της τεχνικής μελέτης και των δοκιμών και των σχετικών εκθέσεων που παρουσιάστηκαν και συζητήθηκαν στην Επιτροπή. Αυτό δεν ήταν όλο, όλη η προσέγγιση. Επίσης, στην εξέταση της όλης ενίας ε, προέβησε σε συζητήσεις με το Συμβούλιο Ευρωπαϊκή Επιτροπή με το Ευρωκοινοβούλιο, με την Επιτροπή σας διοργανώθηκε μια συνάντηση από τη γραμματεία της ΛΥΜΠΕ τον Φεβρουάριο του 2015 στη Δικηβολευτική Επιτροπή για Ατεφή Σύνορα, μεγάλη εκδήλωση ε, που τροφοδότησε τη διαδικασία. Οι υπηρεσίε Ευρωπαϊκής Επιτροπής διενήγησαν διάφορες συζητήσεις τεχνικού περιεχομένου με διάφορα θέματα και συγητές για το πακέτο του 2013. Ο κύριος Ντεμέρα και η κυρία Φαγιόν συμμετείχαν και οι σκιώδεις Είχαμε συγκεκριμένες συναντήσεις με εκπροσώπους ε, του EDPS, της Υπηρεσίας επίσης για θεμελιώδη δικαιώματα, εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών, ε, αστυνομικές αρχές, μεταφορείς κλπ. Έγιναν πολλές συναντήσεις, έγινε και δημόσια διαβούλευση, καλέσαμε πολίτες ε, και από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εκτός Ευρωπαϊκής Ενώσεως να συμμετάσχουν. Ετοιμάσαμε και αξιολόγηση αντικτύπου που υιοθετήθηκε από το ρυθμιστικό φορέα φέτος τον Ιανουάριο και ήταν σημαντικό να πούμε ότι αυτή η εκτίμηση συνεπιών έκανε και αξιολόγηση όσον αφορά τα θεμελιώδη δικαιώματα που εδραζόταν επί της έρευνας που έκανε και η υπηρεσία για τα θεμελιώδη δικαιώματα κατά τη διάρκεια των δοκιμών πέρσι. Όλα αυτά λοιπόν έγιναν. Οπότε η πρόταση του 2016 βασίζεται επί ε, πολύ εμπαριστατωμένων ε, στοιχείων. Πολλοί συμμετείχαν, είναι προτάσει Ευρωπαϊκή Επιτροπή, έγινε όμω μια διεξοδική ε, συνεργασία με συμμετοχή όλων των εμπλεκομένων φορέων. Α δούμε λοιπόν το σύστημα εισόδου-εξόδου. Ε, εν κατακλείδη θα εφαρμόσει υπηκόστη των χωρών και για εκείνου που απαιτείται θεώρηση και για εκείνου που δεν απαιτείται θεώρηση που ε, εισέρχονται για σύντομο χρονικό διάστημα στην, στο χώρο Σέγγεν μέχρι 90 ημέρες. Για επισκέπτες μιλάμε εκτιμήθηκε το 2015 ότι μιλάμε για περίπου 200 εκατομμύρια διαλέψεις των συνόρων Σέγγεν, εισόδου-εξόδου. Το σύστημα εισόδου-εξόδου θα καταχωρεί το όνομα, το ταξιδιωτικό έγγραφο, βιομετρικές πληροφορίες, λεπτομέρειες του ταξιδιωτικού εγγράφου, των υπηκών αυτών. Θα καταχωρείται και θα ε, καταχωρούνται στοιχεία εισόδου-εξόδου. Δηλαδή, τόπο και ημερομηνία εισόδου, τόπο ημερομηνία εξόδου. Το σύστημα αντικαθιστά ε, το σύστημα το χειρονακτικό, το τωρινό και θα συνάδει με την νέα οδηγία την προστασία των δεδομένων και το σχετικό κανονισμό που υθετήθηκαν από το Κοινοβούλιο στις 14 Απριλίου νεστότος έτου. Τι θα δώσει το σύστημα. Καταρχάς, θα δίδονται σαφείς πληροφορίες γρήγορα, αυτομάτως στους ε, ε των συνόρων. Ε, και ε, επίσης και η διάρκεια μπορεί να μείνει ο επισκέπτης. Και επίσης και οι απορρίψεις ετοιμάτων εισόδου θα καταχωρούνται. Θα παρέχεται και υπηρεσία για τους ταξιδιώτες, για τη μέγιστη διάρκεια διαμονής τους που επιτρέπεται. Επίσης θα παρέχει το σύστημα ακριβής πληροφορίες στις μεταναστευτικές αρχές, στις αρμόδιες αρχές και οι πληροφορίες ε, θα αφορούν την άδεια εισόδου στην περιοχή και επίσης ε, θα πρέπει να εντοπίζονται και οι παράτυποι μετανάστες. Θα παρέχονται στοιχεία επίσης στους εκείνους που θεσπίζουν ε, την ομοθεσία για εκείνους που μένουν παραπάνω από το επιτρεπόμενο διάστημα και έτσι ενημερώνονται και αυτοί που διαμορφώνουν την πολιτική θεωρήσεων ταξιδιωτικών θεωρήσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Βασικό στόχο είναι η επιτάχυνση των μεθοριακών ελέγχων όσον αφορά του υπηκοστή των χωρών. Επιτρέπεται αυτόματη διαχείριση των στοιχείων υπό την εποπτεία των ε, μεθοριοφυλάκων. Ε, Αυτοματισμό είναι το βασικό στοιχείο. Και αυτό είναι ένα σύστημα που αντικαθιστά το χειρονακτικό σύστημα με το οποίο βάζουμε τη σφραγίδα στα διαβατήρια. Επίση και οι αστυνομικέ δυνάμει θα έχουν πρόσβαση θα έχουμε ταυτοποίηση των τρομοκρατών, των, των ε, εγκληματιών, θυμάτων, υπόπτων και επίσης θα έχουμε το ιστορικό των του, ταξιδιωτικών κινήσεων των διαφόρων υπόπτων και των θυμάτων και θα συμπληρώνει τα, τις πληροφορίες που βρίσκονται στο σύστημα πληροφοριών Σέγγεν όσον αφορά τις διαφορές σε σχέση με τις προτάσεις του 2013, αναφέρω τις βασικές διαφορές, πρώτη σημαντική διαφορά, είναι η αρχιτεκτονική του συστήματος. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει μόνο ένα σύστημα εισόδου-εξόδου. Δεν θα υπάρξει κεντρικό πρόγραμμα καταχωρήσεως των ταξιδιωτών, αλλά κριτήρια και πρότυπα θα καθορίζονται για τα κράτη-μέλη που θέλουν να έχουν τέτοια στοιχεία σε εθνικό επίπεδο. Άρα η προσέγγιση είναι πιο ευέλικτη εν αυτή τη ενία. δεύτερο, η διαλειτουργικότητα. Κάτι που συζητήθηκε εδώ επανειλημμένα. Θέλουμε να πετύχουμε αποτελεσματικότερη και ταχύτερη διαδικασία στα σύνορα και θα πρέπει να υπάρχει και διασύνδεση με το EAS και με το σύστημα θεωρήσεων των πληροφοριών θα υπάρχει άμεση σύνδεση μεταξύ διαφόρων συστημάτων και έτσι επιταχύνεται η διαδικασία και προστατεύονται και τα δεδομένα. Θα αποφευθεί η ανάγκη επαναλήψεως των δεδομένων. Να βγαίνουν στοιχεία από το VIS και να αποθηκεύεται στο EIS. Τα στοιχεία που είναι στο VIS θα παραμένουν στο VIS. Δεν χρειάζεται λοιπόν να υπάρχει ε, επανάληψη καταχωρήσεως των στοιχείων, Άρα ε, προστατεύεται η ιδιωτικότητα από το σχεδιασμό του συστήματος. Τρίτη σημαντική διαφορά, βιομετρικά στοιχεία. Στην παλιά πρόταση του 2013 είχαμε 10 δαχτυλικά αποτυπώματα. Συζητήθηκε επανειλημμένα αυτό και δεν σας εκπλήσει αυτό. Η αναθερμμένη πρόταση χρησιμοποιεί τέσσερα δαχτυλικά αποτυπώματα και μία εικόνα του προσώπου ε, σαν βασικούς δείκτες ε, ταυτοποίησης. Διευκολύνεται η διέλευση των συνόρων λόγω της εφαρμογής και συστημάτων αυτομάτων ηλεκτρονικών πυλών ο καθένας μπορεί μόνος του να ξεκινά τη διαδικασία διέλυσης συνόρων μόνος του. Πριν φτάσουν ε, στο σταθμό του, που βρίσκεται ο συνοριοφύλακας. Η προστασία των προσωπικών δεδομένων εδώ έχουμε μειώσει αρκετά τον όγκο των προσωπικών στοιχείων που αποθηκεύονται. Το 2013 μιλούσαμε για 36 ομάδες στοιχείων. Τώρα είμαστε στα 26, 26 ομάδες στοιχείων. 26 αρκούν για τη λειτουργία των, του συστήματος. Η περίοδος διατήρησης των στοιχείων. είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αποθηκεύονται τα στοιχεία για 5 έτη, για όλους τους σκοπούς αυτή η διατήρηση των στοιχείων για πενταετία μπορεί να επαναχρησιμοποιηθούν τα στοιχεία για τον ταξιδιώτη. Άμα ήδη έχει δώσει τα στοιχεία του, μπορεί να χρησιμοποιηθούν. Και οι φύλακε των συνόρων μπορούν να προβούν στην αναγκαία ανάλυση κινδύνου. Έχοντα τα στοιχεία στη διάθεσή του για αυτή την περίοδο και, και τα πέντε έτη βασίζονται επίσης και στο μέσο όρο διαρκείας των διαβατηρίων, ισχύω των διαβατηρίων που είναι πενταετής κατά μέσο όρο. Οπότε υπάρξει προσωμείωση του όγκου των στοιχείων με τη διάρκεια των στοιχείων, ισχύω των στοιχείων. Από την αρχή το ΙΕΣ τα κράτη-μέλη μπορούν να έχουν πρόσβαση στις δυνάμεις στο ΙΕΣ ε, υπό συγκεκριμένους όρους ε, όπως έχουν συμφωνήσει και οι άλλα εργαλεία κατά το παρελθόν, για άλλα μέσα, υπό παρόμοιους όρους. Άλλη σημαντική διαφορά είναι το κόστος. Στην πρώτη του 2013, 1,1 δις προβλεπόταν σαν ενδεικτικό ποσό. Μειώθηκε στα 791-793 εκατομμύρια στο απόθεμα που είχαμε προβλέψει. Στους νέους υπολογισμούς με το απουστευμένο αναθερμμένο σύστημα 480 εκατομμύρια ευρώ πιστεύουμε ότι αρκούν για να αναπτυχθεί το σύστημα και για να λειτουργήσει το σύστημα εισόδου-εξόδου. Εντάχει, ο κώδικας φύλαξης συνόρων ε, Σέγγεν, το δεύτερο κομμάτι του πακέτου νομικής φύσεως, εδώ έχουμε προβεί σε τεχνικές αλλαγές, πρέπει να σωματωθούν οι τεχνικές ε, αλλαγές που επιβάλλονται λόγω της αλλαγής του συστήματος. Επικαιροποίηση χρειάζεται. Δύο σημαντικές αλλαγές έχουμε. Μπορεί ο καθένας να, μπορεί να αυτοεξυπηρετούνται οι ταξιδιώτες από τρίτες χώρες. Αυτή η δυνατότητα δεν υπάρχει σήμερα. Μόνο για επικόπου της Ευρωπαϊκής Ενώση υπάρχει. Και δεύτερον, ο κώδικας Σέγγεν πρέπει να προβλέπει νομικό πλαίσιο για τη δημιουργία εθνικών κέντρων εθελοντικές βάσεις δεδομένων μπορούν να δημιουργηθούν αν θέλουν να το κάνουν τα κράτη-μέλη. Μπορώ να πω αυτό κάτι, ίσως κάτι παραπάνω πάνω σε αυτό το θέμα. Η αρχική πρόταση δεν ισχύει πλέον και εξηγούμε στην αξιολόγηση αντιχτύπου γιατί. Υπάρχουν αμφιβολίες όσον αφορά την κρίσιμη μάζα που θα πρέπει να ε, των, των υπηκών τρίτων χωρών που θα θέλουν να εκμεταλλευτούν το σύστημα RTP. Δηλαδή να χρησιμοποιούν το αυτόματο σύστημα. Αν στόχο είναι να διευκολύνουμε αυτόματο σύστημα για να, επιταχύνει η διέλευση, να επιταχυνθεί η διέλευση, τότε η αξία του RTP δεν βοηθά. Δεν πρέπει να έχουμε παράλληλα συστήματα, αν μόνο ωφελούνται λίγοι. Αυτός ήταν ο λόγος που κάνουμε αυτή την αλλαγή και τούτου λεχθέντος, τα κάτι μελη που θα δημιουργήσουμε συστήματα ATP στα πλαίσια διμερών συμφωνιών με προνομιούχες τρίτες χώρες θα μπορούν να το κάνουν αυτό και στο μέλλον βάσει κοινών ε, κανόνων, συμπεφωνημένων κανόνων Σέγγεν. Αυτή είναι η λογική της προσεγγίσεως που ακολουθούμε. Τέλος, επόμενα βήματα. Η πρόταση παρουσιάστηκε στο Συμβούλιο στο Λουξεμβούργο την περασμένη εβδομάδα ασφαλής εσωτερικών, δικαιοσύνη εσωτερικών. Εκφράσαμε την ελπίδα ότι μια συμφωνία μπορεί να επιτευχθεί με τους συνομοθέτες τάχιστα. Στην ανακοίνωση αναφερόμαστε στο τέλος του 2016 και αν συμβεί αυτό, βέβαια αυτό επιτρέπει σε εμά και στο Γιουλίζα να ξεκινήσουν την πρόθεση του συστήματος το 2017 και να λειτουργεί το σύστημα την 1η Πρώτου του 2020. Thank um, Σε ευχαριστώ. Πολύ φιλόδοξο χρονοδιάγραμμα και μεγάλος φόρτος εργασίας. Τώρα θα δώσω το λόγο στον εισηγητή μας, τον κύριο Δίας Δεμέρα, μετά την παρουσίαση που μας έκανε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Στην εισαγωγή σας, κύριε Πρόεδρε, μας εξηγήσετε πολύ εύστοχα το ιστορικό της αποτυχίας αυτού του νομοθετικού σχεδίου, που ευτυχώς ε, το σώσαμε την τελευταία στιγμή, μετά από πολλές εμπειρίες που συγκεντρώσαμε, από τα πιλωτικά προγράμματα και μετά από έντονες συζητήσεις που είχαμε και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και με όλους τους ενδιαφερομένους. Ο κύριος Ρόζενμπορκ Κάτριν και οι σκιώδεις Είμαστε συμπροταγωνιστές σε αυτή την νομοθετική ιστορία. Οπότε, πιστεύω ότι είμαστε σε θέση λόγω των γνώσεων μας και το ότι δεν ξεκινούμε το μηδενός να προχωρήσουμε πολύ πιο γρήγορα αυτή τη στιγμή. Γιατί η νομοθετική πρόταση έχει απλουστευτεί, έχει τελειοποιηθεί και έχει προσαρμοστεί και στο δημοσιονομικό πλαίσιο, γιατί αυτό ήταν ένα από τα προσκόμματα που αντιμετωπίζαμε στην προηγούμενη φάση. Οπότε, στην παρέμβασή μου θα λάβω υπόψη τις δύο προτάσεις αυτή για το σύστημα εισόδου-εξόδου, για την καταχώρηση δεδομένων εισόδου και εξόδου, αλλά και δεδομένων ε, για την άρνηση εισόδου υπηκών τρίτων χωρών που διέρχονται από τα εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και, τις, και τους όρους πρόσβασης στο σύστημα εισόδου-εξόδου. Επίσης θα μιλήσω και για την τροποποίηση του κανονισμού 2016-399 που αφορά το σύστημα εισόδου-εξόδου. Ε, επαναλαμβάνω λοιπόν, χαιρετίζω αυτή την νομοθετική πρόταση που περιλαμβάνει σημαντικά ε, θέματα όπως τον περιορισμό των βιομετρικών αναγοριστικών στοιχείων που είναι περίτα εξασφαλίζει την απαραίτητη διαλειτουργικότητα με το σύστημα των θεωρήσεων, προβλέπει πρόσβαση στο σύστημα των αρχών επιβολής του νόμου, προβλέπει μείωση του προϋπολογισμού που πέρασε από 1,1 δις σε πάνω από γύρω στα 500 εκατομμύρια. Όλα αυτά έδωσαν πολύ μεγάλη και σημαντική προστιθέμενη αξία στο νέο νομοθετικό σχέδιο. Εμείς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα εξετάσουμε ενδελεχώς τη νέα πρόταση και θα βελτιώσουμε κάποιες πτυχές ε, της προστασίας των δεδομένων, ώστε να είναι πλήρως προσαρμοσμένη στην οδηγία της 14 Απριλίου του 2016. Και για την επεξεργασία των βιομετρικών στοιχείων, ευτυχώς περνάμε από τα 10 δακτυλικά αποτυπώματα στα 4 ε, και ε, περιλαμβάνουμε και την αναγνώριση προσώπου, καταργώντας το θέμα της ε, ήριδος του ματιού. Παρόλο που ήταν πλήρης η παρουσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, δεν μίλησε για τη σημασία των επιταχυντών. Γιατί? Για να επιταχύνουμε τις διαδικασίες στα σύνορα, γιατί το κλειδί της νέας νομοθετικής πρότασης είναι κυρίως αυτή η επιτάχυνση των συνοριακών διελεύσεων. Γι' αυτό και το θέμα των επιταχυντών είναι σημαντικό. Επίσης θα εξασφαλίσουμε τη διαλειτουργικότητα με το σύστημα των θεωρήσεων, σύστημα πληροφοριών θεωρήσεων και ε, θα έχουμε μια σύνδεση με τα εθνικά συστήματα εισόδου-εξόδου. Σε ό,τι αφορά το χρονοδιάγραμμα, θα ήθελα να έχουμε κάποιες συνομιλίες ε, με την Προεδρία του Συμβουλίου ε, και το, τον Επίτροπο και μάλιστα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι πολύ πρόθυμη για συνεργασία και την ευχαριστώ θερμά. Έχουμε συναντήσει και με το EU ΛΙΣΑ. Ήδη είχαμε μία και πολλές άλλες διαβουλεύσεις στις προηγούμενες ε, νομοθετικές φάσεις. Θα μιλήσω λοιπόν και με το EU για να μιλήσουμε και την προστασία των δεδομένων, την πρόσβαση των αρχών επιβολής του νόμου στο σύστημα, το θέμα της απλωστευμένης αρχιτεκτονικής του συστήματος Κάπω σχηματικά μας τα παρουσίασε και ο κύριος Ρόζεμπουργκ. εκπρόσωπος Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Θα μιλήσουμε για τη λειτουργικότητα, ε, τις ε, υποδομές, ε, για την επαφή χρειαζόμαστε ένα ασφαλές δίκτυο, χάρη στο οποίο θα μπορούμε να ανταλλάσσουμε πληροφορίες και δεδομένα με τις εθνικές μονάδες και αρχές. Επίσης, τι γίνεται με τις συνέπειε με τις για τους ταξιδιώτες, γιατί θα κατεργηθεί η σφραγίδα στα ταξιδιωτικά έγγραφα. Οπότε θα πρέπει να έχουμε ένα σύστημα για να γνωρίζουμε πότε ε, θα εισέρχεται και θα εξέρχεται από την Ένωση ο ταξιδιώτης. Σε ό,τι αφορά τα βιομετρικά στοιχεία, θα απαιτήσουμε κάποιες προδιαγραφές ποιότητας, γιατί χωρίς τέτοιες προδιαγραφές ποιότητας για τα βιομετρικά στοιχεία δεν θα μπορέσουμε να τα χρησιμοποιήσουμε αποτελεσματικά. Σε ό,τι αφορά την διευκόλυνση και την επιτάχυση στη διέλευση των, των συνοριακών σημείων, πολύ σημαντικό θέμα. Θα έχουμε πολλές τεχνικές συναντήσεις και μία δημόσια ακρόαση για το θέμα αυτό και θα παρουσιάσω με ρεαλισμό το σχέδιο το Σεπτέμβριο. Νωρίτερα δεν γίνεται. Για να είμαστε ρεαλιστές θα πρέπει να τηρήσουμε αυτό το ε, χρονοδιάγραμμα και δεν μπορούμε να τα διεκπαιρεωσουμε αρων αρων γιατί και προσωπικά έχω ένα πρόβλημα, γιατί έχουμε και βουλευτικές εκλογές τον Ιούνιο. Οπότε για να παρουσιάσω μια σοβαρή έκθεση ε, και πλήρη θα χρειαστώ μέχρι και το Σεπτέμβριο. Επίσης είμαστε παλιές καραβάνες μερικοί σε αυτό το θέμα, άλλοι ε, είναι πιο καινούργοι. Πάντως ε, είμαι πρόθυμος και δεκτικός να συνεργαστώ με τους συναδέλφους τους ευχαριστώ θερμά και παραλαμβάνω την ευγνωμοσύνη μου και τα συγχαρητήριά μου και ευχαριστώ θερμά και την Κατρίν που από τη γραμματεία θα προσφέρει ανεκτήμητη βοήθεια γιατί είναι πολύ καλά εξοικειωμένη με την έκθεση αυτή. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Είναι μεγάλο θέμα και ευαίσθητο η προστασία των δεδομένων. Σας ευχαριστώ λοιπόν για το έργο σας. Δύο σκιώδεις έχουμε μαζί μας. Θα τους δώσω το λόγο. Για τους φιλελεύθερους, η κυρία Μέλναρ. Ευχαριστώ πολύ. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Τεμίρες γιατί θεωρούμε ότι η έκθεση βρίσκεται σε καλά χέρια και Περιμένουμε τη συνεργασία μαζί σας. Ε, φυη συνορα σύνορα, σύστημα εισόδου-εξόδου. Ε, πρόκειται για την τέταρτη βάση δεδομένων. Στην ε, ανακοίνωση για τα ευφυή σύνορα, την ασφάλεια και την προστασία, η μεγαλύτερη ανησυχία μας εξακολουθεί να είναι η μη εφαρμογή των υφιστάμενων μέτρων από τα κράτη-μέλη. Ακόμα και στις περιπτώσεις όπου εφαρμόζονται τα μέτρα, η ποιότητα των καταχωρηθέντων ε, δεδομένων δεν ανταποκρίνεται σε απαιτήσει ποιότητα. Γι' αυτό το λόγο το ερώτημα είναι γιατί χρειαζόμαστε μια νέα βάση δεδομένων πριν, πριν γίνει μια ε, ε σε βάθος ε, αξιολόγηση των υφιστάμενων συστημάτων. Επίσης η Europol δεν έχει ακόμα αξιοποιήσει πλήρως τη δυνατότητά της να ε, έχει πρόσβαση στην κεντρική βάση δεδομένων. Η Κομισιόν ε, παρουσίασε κάποιες προτάσεις για τη βελτίωση της διασυνδεσιμότητας και της διαλειτουργικότητας. Στην ανακοίνωση η αξιολόγηση αποκαλύπτει ότι η διαλειτουργικότητα είναι προβληματική και εγώ θα ήθελα να μάθω πώς θα αποτραπεί στο μέλλον ε, πώς αποτελούν τα προβλήματα. Τέλος, το σύστημα εισόδου-εξόδου δεν θα ε, επεκτείνει τις ε, υποχρεώσεις καταγραφής των δεδομένων για όλους τους υπηκόους τρίτων χωρών, ιδιαίτερα αυτούς που ξεπερνούν την άδεια παραμονής τους. Για αυτούς συγκεκριμένα, να πω κάτι. Γιατί χρειαζόμαστε τον αριθμό εκείνων που ξεπερνούν το, την άδεια παραμονής τους. Εντάξει, θα μάθουμε έναν αριθμό, αλλά δεν θα ξέρουμε τι να τους κάνουμε αυτούς του ανθρώπου. Άρα ε, είναι κάτι που τελικά ε, ευνοεί τους ε, λαϊκιστές. Και ως Αυστριακή μπορώ να σας πω από δική μου εμπειρία στη χώρα μου για το τι συμβαίνει όταν δίνουμε επιχειρέματα στους λαϊκιστές. Άρα γιατί θέλουμε να μάθουμε αυτόν τον αριθμό και τι θα τον κάνουμε σε τελική ανάλυση αυτόν τον αριθμό. Ελπίζω ε, να μην πρόκειται άλλη μια φορά για μια βιαστική ε, ε νομοθετική πρωτοβουλία ε, εγώ σε κάθε περίπτωση δεν πιστεύω καθόλου ότι, έχουμε, ότι ακολουθούμε το σωστό δρόμο σε αυτό το θέμα. Ευχαριστώ Σκιώδης για την ε, ε, Γκουε, είναι η κυρία Βέρζια. Ευχαριστώ. Και ευχαριστώ και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την παρουσίαση που μας έκανε, που ήταν ιδιαίτερα μεστή και εμπεριστατωμένη. Και ευχαριστώ και τον εισηγητή μας με τον οποίο συνεργάζομαι με ιδιαίτερη χαρά εδώ και πολλά χρόνια και με ικανοποίηση θα συνεργαστούμε και σε αυτό το ζήτημα. Το, ήδη το ιστορικό τίτλο έκθεση αυτή ε, είναι, προϋποθέτει τεράστιο πρόγραμμα. Τα έξυπνα σύνορα, η διαμόρφωση των ευφυών σύνορων. Τι σημαίνει αυτό. Εντάξει, να δώσουμε έξυπνες πληροφορίες δεν νομίζω ότι ισχύει κάτι τέτοιο. Από την αρχή ε, έχουμε σημαντικές εξέλιξεις. Στην αρχή μας είπαν ότι πρώτα απ' όλα θέλαμε να διευκολύνουμε τη διέλευση των συνόρων. Περί αυτού επρόκειτο στην αρχή. Αλλά τελικά καταλάβαμε ότι το θέμα ήταν η παροχή πληροφοριών και η καταπολέμηση της παράτυπης μετανάστευσης γιατί μας είπαν ότι εξακριβώνουμε την ημερομηνία εισόδου και κυρίως την ημερομηνία εξόδου για να γνωρίζουμε ποιοι βρίσκονται παράτυπα στην Ευρωπαϊκή Επικράτεια. Διαπιστώνω βέβαια ότι έχουμε καμιά δεκαριά νομοθετικά κείμενα και προτάσεις που μελετούμε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που πάνε όλο προς την ίδια Και αρχίζω να τα έχω χαμένα. Νομίζω ότι δημιουργούμε εδώ ένα παραπέτασμα καπνού, δημιουργούμε βάσεις δεδομένων, ε, συστήματα και δεν έχουμε τις ίδιες πληροφορίες σε όλες τις βάσεις δεδομένων. Και θέλουμε και μια διασυνδεσιμότητα. Πολλά λόγια του αέρα μου φαίνονται. Γιατί δεν έχουμε ένα ενιαίο σύστημα, αλλά έχουμε κοινού κανόνες, λέμε. Νομίζω ότι κοροϊδεύουμε του εαυτού μα και του άλλου. Γιατί αν θέλουμε να είμαστε πραγματικά αποτελεσματικοί, χρειαζόμαστε ένα κοινό σύστημα. Γιατί του κοινού κανόνε του ξέρουμε. Τα κράτη-μέλη κάνουν το κεφαλιού του και θα συνεχίσουν να το κάνουν αν δεν έχουμε ένα κοινό σύστημα. Και αυτό ισχύει για την καταπολέμηση τη τρομοκρατία επίση. Γνωρίζουμε ότι το θέμα είναι η συνεργασία. Οπότε τι κάνουμε τελικά. Χαίρομαι που περάσαμε από το 1,1 δις σε 480 εκατομμύρια. Αλλά και 400 εκατομμύρια δεν είναι λίγα. Χαίρομαι που μειώθηκε ο προπολογισμό, αλλά πώς θα δαπανηθούν αυτά τα 400 εκατομμύρια, τι εξυπηρετούν. Έχουμε ένα σωρό άλλες δομές. Επίσης, το θέμα της διασυνδεσιμότητα με απασχολεί κάπως. Ερωτώ λοιπόν. Πώς θα τα εναρμονίσουμε όλα αυτά μακροπρόθεσμα με ένα κείμενο που ε, θα εγκρίνουμε για την ε, εξακρίβωση των ε, κατάλληλων στοιχείων. Δεν θα είναι πια έξυπνα, αλλά κατάλληλα. Και μας είπαν ότι το σύστημα θα υιοθετηθεί, θα, θα εφαρμοστεί το 2020 με την ραγδαία όμως εξέλιξη των τεχνολογιών. Πολύ φοβούμε ότι όταν εφαρμοστούν όλα αυτά το 2020 θα είναι πλέον παροχημένα και θα χρειαστεί να ξαναγυρίσουμε α, στο, στην αρχή. Κάτι που είδαμε και στην περίοδο του συστήματο πληροφοριών για τις θεωρήσεις και του συστήματο πληροφοριών Σέγγεν. Φαίνεται θα να του τους πολίτες. Μην εκπλήστε λοιπόν από τα αποτελέσματα των λαϊκιστών σε ορισμένε χώρε. Γιατί ακριβώς επειδή προσπαθούμε να προλάβουμε τι ακραίε δεξιέ σχέσει, τελικά είναι λογικό οι πολίτες να προτιμούν το πρωτότυπο από το αντίγραφο. Και αυτό πραγματικά με φέρνει σε μια απόγνωση. Ευχαριστώ πολύ. Πρωτού ξαναδώσω το λόγο στον κύριο Δίας Ντεμέρα. Μήπως θα ήθελε το Συμβούλιο να πάρει το λόγο πολύ σύντομα για να μας ενημερώσει. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ τους βουλευτές και μέλη της Επιτροπής. Πράγματι, περιμέναμε πολύ καιρό αυτή την ε, πρόταση στο Συμβούλιο από το 2008. Θεωρούμε ότι πρέπει να εξοχρονιστεί η διαδικασία ελέγχου των συνόρων ε, και τη διαδικασία σφράγισης. Είχαμε τρία χρόνια έντονων συζητήσεων και εδώ στο Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο. Είχαμε ε, μελέτες τεχνικές που αποτέλεσαν και τη βάση για τις νέες προτάσεις. Θεωρούμε ότι οι προτάσεις αυτές είναι αναγκαίες για την καταπολέμηση της παράνομης μετανάστευσης, για την παροχή της δυνατότητας εντοπισμού ανθρώπων που ξεπερνούν την άδεια παραμονής τους, αλλά και για, βεβαίως για την νόμιμη μετανάστευση και για ε, τα ταξίδια. Ε, οι Υπουργοί έχουν συμφωνήσει ότι οι, οι προτινόμενες αλλαγές αποτελούν ένα καλό παράδειγμα διασυνδεσιμότητας. Γι' αυτόν τον λόγο το Συμβούλιο πιστεύει ότι οι προτάσεις της Κομισιόν αποτελούν σωστή βάση και ε, επιθυμεί να ε, καταλήξουμε σε συμφωνία μέχρι το τέλος της χρονιάς. Για το σκοπό αυτό η Προεδρία έχει ξεκινήσει τις εργασίες της για το επί του κειμένου και περιμένουμε να ολοκληρώσουμε αυτή τη βδομάδα την πρώτη ανάγνωση στην ομάδα εργασίας Frontex. Και ελπίζουμε η Προεδρία να καταφέρει να κάνει κάποια σημαντικά βήματα ε, προς το στόχο της, ε, ε, του να καταλήξουμε σε ένα κείμενο. Βρισκόμαστε σε συνεργασία με τον κύριο Ντεμίρα και ε, προσβλέπουμε σε μια επικοδομητική συνεργασία με τον εισηγητή και με τους σκιώδεις συντονιστές του Κοινοβουλίου. Ευχαριστώ. Η Κομισιόν θέλει να κάνει κάποια άλλα σχόλια. Όχι. Κύριε Δίας Ντεμέρα, θέλετε να πάρετε ξανά το λόγο για τις τελικές σας παρατηρήσεις. <coughs> Κύριε Πρόεδρε, αντί για συμπέρασμα και χάρη κοινοβουλευτικής αυρότητας, θα ήθελα να ευχαριστήσω τις κυρίες Μέσνα και Βερζιά για τα σχόλιά τους που θα λάβω πολύ σοβαρά υπόψη. Θεωρώ ότι η γνώση είναι η βάση της συζήτησης αλλά και της κριτικής. Και πιστεύω ότι όταν εμβαθύνομαι από κοινού, και το τονίζω, από κοινού, ε, και εξοικειωθούμε με την νομοθετική πρόταση, τότε θα καταφέρουμε να λιάνουμε τις διαφορές μας και τις αποκλήσεις μας και να μεγιστοποιήσουμε τη σύγκληση και τα κοινά μας σημεία. Και για μένα είναι ιδιαίτερη χαρά η συνεργασία με τις κυρίες αυτές. Το Συμβούλιο μίλησε πολύ καθαρά και με μεγάλη σαφήνεια. Το νομοθετικό αυτό σχέδιο έχει δύο όψεις. Είναι σαν το νόμισμα. Η μία όψη αφορά τη διευκόλυνση της ε, διέλευσης και της νόμιμης ε, ε, διέλευσης των συνόρων και από την άλλη εντοπίζει τις παράτυπες μετακινήσεις. Δεν μπορούμε λοιπόν με λιγότερα λόγια να μιλήσουμε τόσο σαφώς. Χαίρομαι για τη συνεργασία και με το Συμβούλιο και με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και από εδώ και πέρα να σκομπονόμαστε και ξεκινούμε τη δουλειά. Ευχαριστώ κύριε Δεμέρα. Όπως είπαν και άλλοι συνάδελφοι, έχουμε εμπειρία πλέον. Ευχαριστώ και εσάς και τους σκιώδους και υπάρχει και μια ε, ακρόαση που θα γίνει στο ε, το επόμενο διάστημα. Ελπίζω και να συμμετάσχουν μαζικά τα μέλη τη Επιτροπή μα. Μπορούμε να περάσουμε στο επόμενο θέμα, στο σημείο 11 τη ημερήσιας διάταξη. Γενικός Προϋπολογισμός τη Ευρωπαϊκή Ένωση για το οικονομικό Έτο 2017, σε ό,τι αφορά την Επιτροπή μα. Η κυρία Μακοβέη είναι καθοδόν. Περιμένουμε να καταφτάσει. Να σας παρουσιάσω λοιπόν αυτό το θέμα. Με βάση την αιτήσια διαδικασία θα γίνει ανταλλαγή απόψεων με, την, ε, με τους ηγητές της Επιτροπής Προϋπολογισμών για το οικονομικό έτος 2017. Ο διάλογος λοιπόν θα γίνει ως εξής. Πρώτα θα δώσουμε το λόγο στον κύριο Γιένς Κάιερ. Σας καλωσορίζω θα μας προσάσει τις προτεραιότητες και μετά θα έρθει η κυρία Μάκοβε η οποία θα μιλήσει για τις προτεραιότητες της Επιτροπής ΛΥΜΠΕ. Και αν υπάρξει χρόνος θα δώσω το λόγο στους σκιώδεις και στα υπόλοιπα μέλη της Επιτροπής μας. Κύριε Γκάιρ, θα περιμένετε λίγο μέχρι να φτάσει η κυρία Μακοβέ, Δεν έχετε αντίρρηση, έτσι δεν είναι. Μην φεύγετε, συνάδελφοι, η κυρία Μακοβέη έρχεται. This is what happens when you stick to time. We were bang on 10.30. That's always a mistake. Αυτά παθαίνουμε όταν τηρούμε το χρονοδιάγραμμά μας. Είμαστε στην ώρα μας, Ακριβέστατη και συνεπέστατη στις 10.30 και εδώ καθυστέρηση. Jens, maybe, um, we... Jens, ε, ε, μάλλον καλύτερα είναι να ξεκινήσουμε γιατί δεν ξέρουμε πότε ακριβώς θα καταφτάσει η κυρία Μακοβέη. Ε, ας ξεκινήσουμε λοιπόν την συζήτηση εμείς και όταν φτάσει η κυρία Μακοβέη θα της δώσουμε το λόγο. Ο λόγος λοιπόν στον κύριο Γιένς Γκάιερ θα μας παρουσιάσει τις προτεραιότητες της Επιτροπής Προϋπολογισμών. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, σήμερα είναι η, η μέρα που ε, είχε ανακοινωθεί ότι θα ότι θα, ότι θα κοινωθεί αύριο δηλαδή ο, ο Γενικός Προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για αύριο είχε ε, προγραμματιστεί κανονικά τελικά θα αναβληθεί τέσσερις εβδομάδες η διαδικασία αυτή και ο λόγος που ε, ισχυρίζεται η Επιτροπή ότι ε, συνέβη αυτό είναι τα, ότι το γεγονός ότι τα, τα έξοδα και το κόστος της διαχείρισης της προσφυγικής κρίσης δεν έχει ακόμη ε, εκτιμηθεί πλήρως. Ε, φυσικά είναι Απολύτω ε, συμπτωματικό το γεγονό ότι απλά αναβάλλεται η δημοσίευση του προπολογισμού για την περίοδο μετά το δημοψήφισμα. Φυσικά δεν συνδέονται καθόλου ε, αυτά τα δύο ζητήματα. Ε, ηρωνικά βέβαια το λέω. Η αναβολή αυτή, η χρονική, πράγματι είναι αλήθεια ότι δεν περιπλέκει τα πράγματα ιδιαίτερα. Απλά με βάση την ε, εσωτερική μας διαδικασία δεν θα λάβουμε απόφαση ε, σχετικά με την διαπραγμάτευση που θα γίνει με το Συμβούλιο. Δεν έχουμε χρόνο για κάτι τέτοιο. Ε, στην πραγματικότητα όμως οι δυσκολίες αφορούν κυρίως το Συμβούλιο, διότι το Συμβούλιο ε, κάνει πρώτο τις τροποποιήσεις ε, στην πρόταση της Κομισιόν και εμείς σε δεύτερο χρόνο μπαίνουμε στη φάση των διαπραγματεύσεων ως Κοινοβούλιο. Θα υπάρξει λοιπόν μια διαδικασία για την εφαρμογή του προϋπολογισμού, όπως έγινε και το 2014, διότι οι ευρωεκλογές ε, μας ανάγκασαν τότε, εκείνη τη χρονιά, να αναβάλουμε, να αναστείλουμε τις εργασίες μας για έξι εβδομάδες. Θα περιμένουμε και τις ε, γνωμοδοτήσεις των ε, επιτροπών και των τεχνικών τμήματων που θα συνδυαστούν και θα συνεκτιμηθούν με ε, όλες τις υπόλοιπες απόψεις και γνωμοδοτήσεις που θα εκφράσει το Κοινοβούλιο και όλα αυτά στο τέλος θα ε, συνδιαμορφώσουν την θέση του Κοινοβουλίου. Τον ε, Απρίλιο είχαμε εδώ υπερψηφίσει το Κοινοβούλιο, στην Επιτροπή μάλλον Προπολογισμών, με μεγάλη πλειοψηφία τις δικές μας κατευθύνσεις και είχαμε πει ότι ε, οι συνθήκες, ε, ότι οι γενικές συνθήκες δεν αλλάζουν από τη σκοπιά του προϋπολογισμού τουλάχιστον μέσα σε ένα διάστημα 12 μηνών. Η Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων και η Επιτροπή Προϋπολογισμών έχει ασχοληθεί με την προσφυγική κρίση και δεν χρειάζεται εδώ να σας πω πόσο μεγάλες ήταν οι δημοσιονομικές και οικονομικές προκλήσεις που δημιούργησε αυτή η προσφυγική κρίση. Αυτή τη στιγμή έχω πολύ μικρές ελπίδες ότι οι προκλήσεις αυτές για το 2017 θα είναι πολύ διαφορετικές από ό,τι ήταν για φέτος. Και αυτό είναι σημαντικό γιατί στην κατηγορία, τη δημοσιονομική κατηγορία 3, ε, όπου εμπίπτουν τα ταμεία και τα κονδύλια με τα οποία ασκείται και υλοποιείται η πολιτική, έχουν εξαντληθεί πλήρως. Και στην πραγματικότητα μόνο το, το μέσο ευελιξίας του προϋπολογισμού εξασφαλίζει την ε, πρόσβαση και την συμμετοχή του Κοινοβουλίου, μέσω, του οποίου, μέσω της οποίας ε, ε, διαδικασίας καταφέραμε να παρέμβουμε και να ανταποκριθούμε στις ε, ανάγκες που προέκυψαν. Εγώ δεν ε, θεωρώ ότι είναι πιθανό να εξαντληθούν για άλλη μια φορά τα κονδύλια της κατηγορίας 3. Με άλλα λόγια δηλαδή αυτό που θέλω να πω είναι ότι θα έχουμε πολύ μικρά οικονομικά και δημοσιονομικά περιθώρια για τη χρηματοδότηση όλων των αναγκών. Και το λέω με πικρία αυτό, διότι τα κράτη-μέλη ήταν εκείνα που είχαν επενέσει το ένα το άλλο το 2013 όπως είπα για το ότι πρόκειται για τον πρώτο ε, προϋπολογισμό που μειώνεται. Και τώρα ερχόμαστε και διαπιστώνουμε ότι αυτό το μεσοπρόθεσμο δημοσιονομικό πρόγραμμα ήταν τελικά ένας προϋπολογισμός που δεν αντεποκρινόταν ε, ή δεν μπορούσε, δεν ήταν έτοιμος να αντεποκριθεί σε όλες τις συνθήκες. Φαίνεται τώρα, λόγω της κρίσης, ότι τελικά δεν ε, ήταν επαρκής ο προϋπολογισμός αυτός. Αυτή είναι η βάση και η σκοπιά, το πρίσμα μέσα από το οποίο θα πρέπει να ε, εξετάσουμε τις ε, διαπραγματεύσεις για τον προϋπολογισμό που έχουμε μπροστά μας. Μέχρι το φθινόπωρο περιμένουμε και μια πρόταση αναθεώρησης του πολιτού δημοσιονομικού πλαισίου. Εμείς μιλούμε δηλαδή για αναθεώρηση. Τα κράτη-μέλη μιλούν πιο πολύ για ένα review Το Κοινοβούλιο όμως έχει σαφή άποψη ότι χρειάζεται ριζική αναθεώρηση γιατί ακριβώς τα κονδύλια δεν φτάνουν. Δεν είναι βέβαια το μόνο πρόβλημα. Η κρίση εξακολουθεί να σοβεί, η οικονομική κρίση σε διάφορες ε, χώρες. Χρειάστηκε να βρούμε 3 δισεκατομμύρια για να μπορέσουμε να χρηματοδοτήσουμε επαρκώς το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων και όλα αυτά με την ταυτόχρονη υποχρέωση να λαμβάνονται υπόψη και οι προτεραιότητες της στρατηγικής Ευρώπη 2020 και αναφέρομαι συγκεκριμένα στις ε, προτεραιότητες και στις πρωτοβουλίες για την καταπολέμηση ε, της ε, φτώχειας, της ανεργίας των νέων. Σε αυτή τη βάση λοιπόν αποφασίσαμε ότι στις κατευθυντήρες γραμμές θα πρέπει τα διάφορα οικονομικά εργαλεία που θέτει στη διάθεσή μας η Κομισιόν για να αναλύσει την οικονομική κατάσταση. Να συνδεθούν λοιπόν αυτά τα εργαλεία με, στενότερα δηλαδή με τον προϋπολογισμό. Έχουμε έκθεση για την ανάπτυξη, έχουμε ευρωπαϊκό εξάμεινο. Είναι όλα αυτά μέσα και εργαλεία που καταδεικνύουν τι μπορούν να κάνουν τα κράτη-μέλη προκειμένου να ε, ενισχύσουν την ε, οικονομική τους ευρωστία και την ανταγωνιστικότητα τους αλλά εμείς θεωρούμε ότι αν συνδεθούν αυτά τα εργαλεία πιο στενά με τον προϋπολογισμό, θα αυξηθεί και η προστιθέμενη ευρωπαϊκή αξία. Αυτή λοιπόν είναι η βάση ε, της δικής μας στάσης και προσέγγισης Και να πω ότι παρά το γεγονός ότι αναβλήθηκε η διαδικασία η δημοσίευση του προπολογισμού τέσσερι εβδομάδε, εξακολουθούμε να είμαστε υποχρεωμένοι να τελειώσουμε τη διαδικασία αυτή στο τέλος χρονιάς. Αυτά ήθελα να σας πω εγώ από τη δική μας πλευρά, για να σας περιγράψω ποια είναι η γνώμη τη Επιτροπής Προπολογισμών για την συζήτηση που έχει ξεκινήσει και με ποιε βασικέ αρχέ ε, προσερχόμαστε εμεί στη συζήτηση. Το Συμβούλιο τώρα έχει, έχει χωριστεί σε τρία τμήματα. Ε, οι φίλοι των αγροτών, οι φίλοι της συνοχής και οι φίλοι των εκπτώσεων. Και το όλο θέμα της συζήτησης ε, είναι βεβαίως πόσα χρήματα θέλουν τα κράτη-μέλη να διαθέσουν ε, στον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και εδώ το κύριο ζήτημα αφορά βεβαίως τις, πληρωμέ. πληρωμές. Και εδώ το, θέμα που ε, τους αφορά πολιτικά, τα κονδύλια της κατηγορίας 3, 3 δεν θα τους δώσει τη δυνατότητα να ε, ε κάνουν μεγάλες ε, τροποποιήσεις. Θα δούμε όμως ότι θα προσπαθήσει το Συμβούλιο το στις άλλες κατηγορίες να γίνουν μεγάλες περικοπές. Αυτά νομίζω είναι τα προβλήματα που θεωρώ ότι θα αντιμετωπίσουμε και είμαι στη διάθεσή σας ε, και περιμένω να ακούσω και τις δικές σας παρατηρήσεις. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ Γιένς. Ήταν ειλικρινής και ανοιχτή αξιολόγηση από πλευράς Επιτροπής Προπολογισμών. Η κυρία Μακοβέη τώρα θα τονίσει τις προτεραιότητε τη Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών όσον αφορά τον προπολογισμό. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ όλους σας για τη δυνατότητα που μου δίνετε για την ανταλλαγή απόψεων. Να υπογραμμίσω κάποια πράγματα θα ήθελα. Καταρχάς πιστεύω ότι περαιτέρω ανακατανομή για κονδύλια που δεν έχουν χρησιμοποιηθεί επαρκώς ή καλά θα πρέπει να εξεταστούν πριν αυξηθούν οι αδίποτε κονδύλια όπου παίρνουμε χάρη με την κατάσταση των προσφύγων. Οι πόροι για το τέλος του 2016 και το πρόγραμμα το αρχικό για το 2017 θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν για τις προσπάθειες μετεγκαταστάσεις που καταβάλουν τα κράτη-μέλη ούτως ώστε να ξαναγεμίσει το Ταμείο για τη μετεγκατάσταση και μετανάστευση διότι έχει εξαντληθεί και πρέπει να στηρίξουμε και την δημιουργία του κονδυλίου που θα χρηματοδοτεί έκτακτη υποστήριξη αυτών των ανθρώπων του ενώσεως με συγκεκριμένη στόχευση. Είναι καλή συμπερίληψη στον προπολογισμό του 2017 των επαρκών πόρων για την υποστήριξη της μετατροπής ε, της Frontex σε μια ευρωπαϊκή ακτοφυλακή και της ΕΑΣΟ σε μια υπηρεσία αρμόδια για το άσυλο. Πρέπει να κάνουμε σωστές επιλογές. ούτω ώστε να εξαιρεθούν οι φορείς που ασχολούνται με τη μετανάστευση από το στόχο του 5% που έχουμε θέσει. Τρίτον, θα πρέπει τα κονδύλια για Europol και Eurojust να αυξηθούν καταλήλως για να διευκολυνθεί η συνεργασία αστυνομικών δυνάμεων και των μυστικών υπηρεσιών για να συντονιστεί η έρευνα που ασκούν όσον αφορά την αντιμετώπιση των τρομοκρατικών απειλών. Το πακέτο για τα φύση σύνορα είναι καλό βήμα πρόοδου. Και το Ευρωπαϊκό Θεματολόγιο για την ασφάλεια και τη μετανάστευση στηρίζονται με αυτόν τον τρόπο και χρειάζεται σωστή χρηματοδότηση για τα φύση σύνορα. Τέταρτον. Εν ονόματι καλώ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μας εξηγήσει λεπτομερώς οι πόροι για τον προπολογισμό του 2017 πώς έχουν υπολογιστεί, θα ήθελα να δω δημοσίευση του πλήρους καταλόγου των αποδεκτών των πόρων. Θα πρέπει να γίνεται τακτική αξιολόγηση της χρήσης των πόρων. Όπως και στις περιπτώσεις και τις περιοχές που δέχονται κατεπίγουσα βοήθεια. Θα πρέπει να γνωρίζει ο κόσμος πώς χρησιμοποιούνται τα χρήματα. Πρέπει να γίνει αξιολόγηση συνεπειών τακτικά. να δούμε πώς η υποστήριξη που παρέχεται κάνει τη διαφορά. Εάν κάνει τη διαφορά. Πέμπτον. Να επιστήσει την προσοχή στο εξή. Μέχρι 2 Ιουνίου είναι στο τόσο η οδήποτε ομάδα ή μέλος επιτροπής που υποβάλει προτάσεις για νέα πιλωτικά προγράμματα και προπαρασκευαστικές δράσεις και προτάσεις για παράταση ισχυών των προγραμμάτων προ αξιολόγηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το αναφέρω αυτό διότι Ίσως κάποιοι συνάδελφοι θα έπρεπε να θυμηθούν ότι υπάρχει αυτή η δυνατότητα και αυτό σχετίζεται με την κρίση την προσφυγική. Αυτά και σας ευχαριστώ. Καλώς. Θέλω να ελέγξω αν κάποιος άλλος θέλει το λόγο. Όχι. Κυρία Σίμπελ και κυρία Σπινέλη. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Σύντομα να προσθέσω κάτι, ένα ή δύο στοιχεία στα υποθέντα αυτά που είπαν οι δύο εισηγητές. Καταρχάς, βέβαια, τις καλές ημέρες που περνάει η κοινωνία μας, ίσως να μην χρειάζονται τα χρήματα, αλλά όταν περνάμε κρίση, πρέπει να αυξάνονται οι προσπάθειες για την αντιμετώπιση των προβλημάτων. Οπότε, είτε θα πάρουμε νέα χρήματα, συμπληρωματικά χρήματα που θα μπουν στον προπολογισμό, είτε για το μέλλον θα πρέπει να αλλάξουμε τους κανόνες για τον προπολογισμό μας. Να μην επιστρέφονται όλα τα μη δαπανηθέντα ποσά, αλλά να παραμένουν τα ποσά αυτά, ούτω ώστε να υπάρχουν κάποια χρήματα στα κονδύλια για περίοδο κρίσεως. Δεύτερον, αυτό χρειάζεται ακόμα περισσότερο, διότι κατανοούμε τώρα ότι κάποια κράτη-μέλη δεν είναι έτοιμα από μόνα τους να συμβάλλουν στην αντιμετώπιση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουμε, όχι την υποστήριξη άλλων χωρών, αλλά δεν, όχι μόνο δεν στηρίζουν άλλες χώρες, αλλά δεν επομίζονται τις δικές τους ευθύνες. Οπότε χρειάζεται μεγαλύτερη ανάληψη ευθυνών α, στον οικονομικό τομέα, στα πλαίσια του προπολογισμού του ευρωπαϊκού. Και κάτι άλλο. Δεν χρειάζονται μόνο περισσότερες προσπάθειες για να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα, τα προσφυγικά, αλλά αν δούμε τις κοινωνίες μας θα δούμε ότι περισσότερες προσπάθειες θα πρέπει να γίνουν για να αντιμετωπιστεί η αύξηση της φτώχειας που ε, χτυπά κάποια κομμάτια, κάποιες, ε, κάποια στρώματα των κοινωνιών μας. Δεν πρέπει να το λησμόνουμε. Ευχαριστώ ε, Μπριγκίτ, η Μπάρμπαρα Σπινέλη. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Εγώ θα ήθελα τέσσερα σημεία να υπογραμμίσω. Το πρώτο είναι η γνωμοδότηση περσινή που ζητούσε δέσμευση για, το, για την έρευνα και διάσωση, πόρους για το Search and Rescue, για να ενισχυθούν οι επιχειρήσεις οι σχετικές των κρατών μελών. Αλλά το κονδύλιο του προπολογισμού, η γραμμή αυτή του προπολογισμού δεν δημιουργήθηκε ποτέ. Δεν ξέρω αν πρέπει να επαναπροταθεί. δεύτερη πρόταση. Η χρηματοδότηση των εθελοντικών δράσεων και της βοηθείας που παρέχεται συγγνώμη, στους ε, πρόσφυγες. Μια, με μια βολιδοσκόπηση που έκανε η Διεθνής Αμνηστία βλέπουμε ότι το βασικό πόρισμα είναι ότι υπάρχει ανοιχτή τοποθέτηση των πληθυσμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά την υποδοχή των προσφύγων κυρίως ε, σε κάποιες χώρες όπως είναι ε, η Βρετανία και η Γαλλία. Τρίτον, η νομική αρρωγή προς τους πρόσφυγες που προσφεύγουν σε αυτή για να μην επαναπατριστούν και τελευταίο σημείο, κατά την άποψή μου ουσιαστικό, η ένταξή τους στην αγορά εργασίας αυτό θα μπορούσε να συνεπιφέρει μια οικονομική ε, συνεισφορά ε, προς τα κράτη-μέλη από πλευράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης για αυτό το σκοπό. Αυτά λοιπόν και σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ Μπάρμπαρα. Δεν θέλει άλλο το λόγο. Οπότε θα ζητήσω τον κύριο Κέρ να δώσει απαντήσεις στα ερωτήματα. Ευχαριστώ. Είμαστε στο ίδιο μήκο από άποψη περιεχομένου. Καμία διαφωνία. Απλά να σας δώσω δύο πληροφορίες όσον αφορά τις ε, παρατηρήσεις της κυρίας Μακοβέη και της κυρίας Σπινέλη. Εγώ δεν είμαι εισηγητής μόνο για, το, για τον προϋπολογισμό 2017, αλλά είμαι και μόνιμος εισηγητής για τους οργανισμούς. Το ερώτημα λοιπόν της χρηματοδότησης και της τελέχωσης των οργανισμών είναι ένα θέμα που με απασχολεί πολύ. Και εγώ υποστηρίζω το αίτημα ο στόχος για μείωση 5% του προσωπικού των οργανισμών να εξαιρεθεί. Και όχι μόνο αυτό. Ε, θεωρώ ότι συνολικά η μείωση του προσωπικού της Κομισιόν ε, είναι ανοησία. Είχαμε συμφωνήσει πριν από μερικά χρόνια να ε, μειωθεί το προσωπικό όλων των οργάνων και των οργανισμών κατά 5%. Όμως η Κομισιόν δεν εξέτασε ναι, δεν, δεν, δεν, δεν συγκέντρωσε όλους τους υπαλλήλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αντιθέτως, επέβαλε αυτό το στόχο για 5% σε, για κάθε έναν οργανισμό ξεχωριστά. Και εκεί όπου, για παράδειγμα, χρειάζεται να αυξηθεί το προσωπικό, όπως είναι η, η, η Frontex, χρειάστηκε να ε, ε, αντληθούν θέσεις προσωπικού από άλλους οργανισμούς. Άρα κάποιοι οργανισμοί έχουν αναγκαστεί να μειώσουν το προσωπικό τους μέχρι και κατά 10% προκειμένου να ε, βρεθούν αυτές οι θέσεις για κάποιες άλλες υπηρεσίες και κάποιους άλλους οργανισμούς. Δυστυχώς στη διαμάχη αυτή ιτηθήκαμε και σε διοργανική συνάντηση που είχαμε με το Συμβούλιο είχαμε συζητήσει το θέμα αυτό, διότι είχαμε την εντύπωση ότι και το Συμβούλιο πρώτα και κύρια δεν θα μπορούσε να συμφωνεί με αυτήν την ε, ε, πρακτική της Κομισιόν. Και μας, μας ξάφνιασε το γεγονός ότι το Συμβούλιο τελικά θεωρεί ότι με τον προπολογισμό του 2004 έχουμε αποδεχθεί αυτόν τον στόχο. Αυτή είναι η κατάσταση. Δεν μας αρέσει, ούτε σε μένα προσωπικά αρέσει, αλλά θεωρώ ότι θα πρέπει να εξαιρεθούν πλέον ε, εγώ θεωρώ ότι πρέπει να εξαιρεθούν, θα έπρεπε κανονικά να εξαιρεθούν οι οργανισμοί από αυτόν τον στόχο του 5% μείωση του προσωπικού, αλλά δυστυχώς χάσαμε. Ιτηθήκαμε και όπως είπα αυτός ο στόχος σημαίνει ότι σε κάποιους οργανισμούς χρειάζεται ή έχουν έχουν ήδη γίνει πάρα πολύ μειώσεις προσωπικών. προσωπικού. Αυτή είναι η συνολική εικόνα και δεν θα πρέπει να τη χάσουμε από τον προσανατολισμό μας. Γιατί θα πρέπει να θυμόμαστε ότι όποτε αποφασίζεται αύξηση του προσωπικού σε κάποιον οργανισμό, αυτό σημαίνει ότι θα γίνεται ακόμα μεγαλύτερη μείωση σε κάποιον άλλον. Και οι αποφάσεις της Επιτροπής ΛΥΜΠΕ ε, μας δημιουργούν, μας στην Επιτροπή Προπολογισμών κάποια προβλήματα και κάποιες δυσκολίες. Τι θέλω να πω. Καταλαβαίνω ότι η ΛΥΜΠΕ θέλει να γνωρίζει πόσα χρήματα διατίθενται για την αναζήτηση και τη διάσωση. Και να ξέρουμε πόσα χρήματα τελικά ξοδεύει η Ευρωπαϊκή Ένωση για αυτόν τον καθόλου σωστό στόχο. Από την άλλη πλευρά όμως, το να δημιουργηθεί μια γραμμή στον προϋπολογισμό σημαίνει πάντοτε ότι χάνουμε και ένα κομμάτι της ευελιξίας μας. Γιατί αυτό σημαίνει ότι η Frontex και η Κομισιόν Εφόσον υπάρχει, ας πάρουμε αυτό το search and rescue, την αναζήτηση και διάσωση. Όποτε αυτό το κονδύλι εξαντλείται, η Κομισιόν και η Frontex μπορούν να πάρουν χρήματα από κάποια άλλη γραμμή για να ενισχύσουν την αναζήτηση και τη διάτωση. Αυτό που θέλουμε να κάνουμε δηλαδή πολιτικά. Αν όμως η γραμμή είναι κενή, τότε απαιτείται να ακολουθήσουμε μια τεράστια γραφειοκρατική διαδικασία για να εξευρεθούν τα απαραίτητα χρήματα. Από απόψη περιεχομένου δεν διαφωνούμε καθόλου, αλλά θέλω απλά να επισημάνω ότι το να καταρτιστεί και να δημιουργηθεί μια γραμμή στον προϋπολογισμό νέα, βεβαίως ενισχύει την διαφάνεια αφενός, ωστόσο τελικά η εξέβρεση των ε, απαραίτητων κονδυλίων όταν εξεντλείται κάποια γραμμή γίνεται αφάνταστα πιο περίπλοκη. Αυτό θέλω απλά να σας πω. Βεβαίως συμφωνούμε, υπάρχει αυτό το πολιτικό υπόβαθρο που το γνωρίζουμε και καταλαβαίνουμε απολύτως ποιο είναι το σκεπτικό του αιτήματό σας. Αλλά θέλω να σας επισημάνω ότι δεν είναι σίγουρο, δεν είναι βέβαιο ότι εξυπηρετείτε κι εσείς πολιτικά τον στόχο που έχετε θέσει και νομίζω ότι αξίζει να το επισημάνω αυτό για να το γνωρίζετε κι εσείς γιατί ο πολιτικός μας στόχος τελικά από την δική σας στάση μάλλον δεν εξυπηρετείται. Thank you very much, Σας ευχαριστώ για όλα όσα μας μεταφέρατε από την Επιτροπή Προϋπολογισμών. Έχουμε ακόμη δύο σημεία πριν τις ψηφοφορίες. Δεν μας μένει και πολλούς χρόνους. Κυρία Μακοβέα, θέλω το λόγο παρακαλώ πολύ σύντομα. Επιγραμματικά. Όχι, ωραία. Ευχαριστώ. Ήταν πολύ χρήσιμη συζήτηση και πολύ σημαντικό το θέμα για μας. Υπάρχουν μερικές διαφορές μεταξύ μας, αλλά είναι ευνόητες, γιατί Έχουμε κάποια κρίσιμα σημεία ως Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών στον προπολογισμό, αλλά η συνεργασία μας είναι πολύτιμη και θέλουμε να συνεχιστεί και καλό θα ήταν να κρατήσουμε τις σχέσεις μας ε, καλές, ε, γιατί είναι ευαίσθητη και θέλουμε έναν σωστό προϋπολογισμό. Ευχαριστώ. Παίρναμε στο επόμενο θέμα, το σημείο 12, την καταπολέμηση της διαφθοράς και συνέχεια στο ψήφισμα της Ειδική Επιτροπής ΚΡΙΜ. Εν είδη και για να σας φρεσκάρω τη μνήμη, με το ψήφισμα της 23ης Οκτωβρίου για την Ειδική Επιτροπή και τα συμπεράσματα της ΚΡΙΜ θα πρέπει να αναλυθούν κάποιες πρωτοβουλίες. Αναθέσαμε στην Επιτροπή ΛΥΜΠΕ ε, να φροντίσει ώστε οι συστάσεις του ψηφίσματος να εφαρμοστούν σωστά σε διοργανικό επίπεδο με βάση αυτές τις στάσεις ε, εκπονούμε μια έκθεση πρωτοβουλίας για την καταπολέμηση της διαφθοράς και τη συνέχεια που πρέπει να δοθεί στο ψήφισμα της Ειδικής Επιτροπής ΚΡΙΜ. Μετά ένα σημαντικό προπαρασκευαστικό έργο καθώς και τη σύνταξη του εγγράφου εργασίας ε, και οργάνωση μιας δημόσιας ακρόασης, ε, παρουσίαση μελετών εμπειρογνωμόνων, ευρωτηματολόγια προς τη Eurojust και τα μέλη από τα κράτη-μέλη Επίσης, ε, ακρόαση με την ε, Ιταλική Επιτροπή κατά τη Μαφία, ε, Είμαστε σε καλή φάση των εργασιών και θα δώσω το λόγο στην εισηγήτρια την κυρία Φεράρα για να μας παρουσιάσει την έκθεσή της. Ευχαριστώ Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω τους κοιόδης ηγητές και το προσωπικό για την πολύτιμη συνεισφορά τους στην σύνταξη του εγγράφου που εξετάζουμε σήμερα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω επίσης και την Γραμματεία της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών για τη θεσιμότητά της, τεχνική υποστήριξη και εκείνους που συμμετείχαν στην ακρόαση που έδωσαν και διάφορες άλλες σκέψεις να λάβουν υπόψη χθες είναι η επέτειο του του Τζοβάνι Φαλκόνε, του, που καταπολέμησε και σε διεθνέ επίπεδο ακόμα τη μαφία, σκοτώθηκε με τη γυναίκα του και του ανθρώπου ασφαλείας του στι 23 Μαου του 1992. Είναι πάρα πολλοί άντρε και γυναίκε που θυσίασαν τη ζωή του στην προσπάθεια καταπολέμησης του οργανωμένου εγκλήματος και για να τονώσουν την νομιμότητα. Θα πρέπει να πούμε ότι θυσίες θυσίε τόσων, ζώων θα παραμείνουν μάτες όσο οι οργανώσεις τύπου μαφίας ε, ελήψη κοινών προδιαγραφών εξακολουθούν θεωρούνται ένα φαινόμενο που αφορά μόνο εθνικά επίπεδα και μπορούν να έχουν ποικίλε δραστηριότητε και να δρούν ταυτόχρονα σε πολλές αγορές, να εκμεταλλεύονται τις διαφορές, ε, τις νομοθεσίες ε, που υπάρχουν μεταξύ κρατών μελών, ούτως ώστε να επεκτείνονται και να μεγιστοποιούν τα έσοδά τους. Το σχέδιο εκθέσεως για την καταβολέμηση της διαφθοράς μετά το ψήφισμα στην Επιτροπή ΚΡΙΜ είναι ένα πρωτοβήμα προς αυτή την, σε αυτή τη θητεία, δηλαδή θα πρέπει να λάβουμε υπόψη το περιεχόμενο και τις στάσεις του ψηφίσματος 23 Οκτωβρίου του 2013 όσον αφορά το οργανωμένο έγκλημα, τη διαφθορά και την ανακύκλωση του χρήματος. Θα πρέπει να εστιαστεί η προσοχή μας επί συγκεκριμένων παρεμβάσεων που έχουν προτεραιότητα ε, θα πρέπει λοιπόν να διτυπώνονται διάφορε προτάσει για την ενίσχυση των δράσεων ε, πολέμηση του οργανωμένου εγκλήματο και τη διαφθορά. Στην αρχική στην αρχική φάση αναφερόμαστε στον έλεγχο και την εφαρμογή των υφεσταμένων νομοθεσιών και την εξολόγηση αποτελεσματικότητα των μέτρων. Αφετηρία της δράση είναι η, η, εφαρμογή από τον κάτω μέλλον των υφισταμένων ε, μέσων που έχουμε σε διεθνέ επίπεδο και επίπεδο Ευρωπαϊκή Ενώση για την κατανάλωση του οργανωμένου κλίματο, ε, τη ανακύκλωση του χρήματο και τη διαφθορά. Σε αυτό το πλαίσιο συστήνεται η προσχώρηση του Ευρωπαϊκή Ενίσου στο Κρέκο ε, που για, μια, για να γίνονται καλύτερα έρευνε. Είναι περίπλοκο λοιπόν αυτό το φαινόμενο και θα πρέπει ο πολιτικός κόσμος να κινηθεί για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος και θα πρέπει, ε, ε όχι, θα πρέπει να καταπολεμηθούμε τα οργανωμένες ομάδες και θα πρέπει να καταπολεμηθεί επίσης και η κύκλωση, το ξέπλυμα του χρήματος. Θα πρέπει να δούμε ότι οι θεσμοί είναι έφραυστοι και ότι δεν μπορούν να κινηθούν επαρκώς για να ανταποκριθούν στην, στις προσδοκίες των πολιτών για την καταπολέμηση αυτών των οργανώσεων και είναι κάτι που διευκολύνει τι εγκληματικέ οργανώσει. Θα πρέπει λοιπόν οι προτεραιότητε για την καταπολέμηση των φαινομένων να πρέπει να καθοριστούν σε συσχετισμό με τι ε, πολιτικέ και οικονομικέ πτυχέ, κοινωνικέ πτυχέ, πτυχέ απασχόληση και παιδεία και εκπαίδευση. Λοιπόν, από επιχειρησιακό επίπεδο, το σχέδιο προτείνει τη δημιουργία μια μονάδα τη Ευρωπόλ ειδική για να καταπολεμά το οργανωμένο έγκλημα και τι ομάδε αυτέ που κινούνται ταυτόχρονα σε διάφορου τομεί και τα κράτη-μέλη θα πρέπει να έχουν ένα όργανο που εξασφαλίζει συντονισμένη δραστηριοποίηση ερευνητική όσον αφορά το οργανωμένο έγκλημα. Όσον αφορά τώρα το νομοθετικό πλαίσιο, κινούμεθα προς ενίσχυση αυτού ζητώντα επεξεργασία ελάχιστων προδιαγραφών και νόμων όσον αφορά τον καθορισμό των εγκλημάτων και το, όσον αφορά το οργανωμένο έγκλημα και τη διαφθορά για να βελτιώσουμε τη συνεργασία τη δικαστική σε διασυνοριακό επίπεδο. Ιδιαίτερη προσοχή δόθηκε μετά στον ορισμό των κοινό του οργανωμένου εγκλήματο και του δημόσιου α, λειτουργού και όσον αφορά του ε, πληροφοριοδότε, θα πρέπει να προστατεύονται επαρκώ. Θα πρέπει να υπάρχει ευρωπαϊκή συγγελία που θα είναι ε, ανεξάρτητη και θα έχει την αναγκαία εξουσία που θα καθορίζεται επαρκώ. Και θα πρέπει να υπάρχει δικαστική αστυνομική συνεργασία που θα είναι ε, η σωστή σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Θα πρέπει να υπάρχει διασυνοριακή συνεργασία αστυνομικών δυνάμεων και δικαστικών φορέων και θα πρέπει να μην έχουμε μακρε διαδικασίε και να μειωθεί η γραφειοκρατία διότι αυτό εμποδίζει την αποτελεσματική καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματο σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Σε αυτό το πλαίσιο ζητείται από τα κράτη-μέλη να αυξήσουν του πόρου που δίδονται για τη συνεργασία των αστυνομικών και δικαστικών αρχών, θα γιάται την αμοιβαία αποδοχή των αποδείξεων, καλείται, οι ερευνητικέ κοινέ ομάδε που χρησιμοποιούνται καλύτερα, θα πρέπει να υπάρχει κοινό σύστημα επικοινωνιών και ανταλλαγή πληροφοριών. Σημασία έχει η στρατηγική που θα πρέπει να ακολουθηθεί όσον αφορά τη εδρομή του χρήματο για να ερευνούνται τα δίκτυα που υπάρχουν το οργανωμένου εγκλήματο και το φαινόμενο τη διαφθορά. Χρειάζεται να ενισχύσουμε τη νομοθεσία και τι διατάξει που θα εγγυώνται μεγαλύτερη διαφάνεια και ανιχνευσιμότητα τη ροή του χρήματο. Πιο συγκεκριμένα στα πλαίσια των Ευρωπαϊκών ε, Ταμείων και Πόρων χρειάζεται τελική επαλήθευση όσον αφορά τη σωστή χρήση των πόρων που διατίθενται. Ιδιαίτερη σημασία έχει η ενίσχυση των μέτρων όσον αφορά την, το πάγωμα και την κατάσχεση των προϊόντων του εγκλήματος και η διασχήριση αυτών των παγωμένων πόρων και των ε, κατασχεθέντων ε, στοιχείων των περισσιακών. Ε, έτσι μπορούμε να εμποδίσουμε τη δύση του οργανωμένου εγκλήματος στην νόμιμη οικονομία. Η διαφθορά είναι ένα από τα βασικά εργαλεία που χρησιμοποιεί το οργανωμένο έγκλημα για να δυσδύσει την νόμιμη οικονομία και να επηρεάσει τι διαδικασίε, τι πολιτικέ, θεσμικέ και τι αποφάσεων και τα κοινωνικά συστήματα των κρατών μελών. Θα πρέπει. Ε, ε υπάρχει παρέκκληση ε, των δημοσίων πόρων ε, και παραποιείται έτσι και ο σωστός ανταγωνισμός. Ζητούμε πιο συγκεκριμένα να ληφθούν μέτρα που αφορούν τους δημόσιους διαγωνισμούς και θα πρέπει να υπάρχει ένα σύστημα, ε, σύστημα ηλεκτρονικών τέτοιων διαγωνισμών για να μειωθεί ε, τελικά το φαινόμενο της διαφθοράς. Τα κρατη πρέπει να εφαρμόζουν συστήματα ε, παρακολούθηση των δημοσίων αυτοδιαγωνισμών και κάθε επιχείρηση που έχει διασύνδεση με οργανωμένο έγκλημα θα πρέπει να αποκλείεται με κάθε οικονομική σχέση με, δημόσιο, με το δημόσιο τομέα. Ένα μέσο που θα πρέπει να εισαχθεί στα κράτη-μέλη ε, είναι μια πιστοποίηση όσον αφορά την ε, μη σχέση ε, μια επιχείρηση με το οργανωμένο έγκλημα και θα πρέπει να ενημερώνεται δόντος και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Όσον αφορά τις παρεμβάσεις, όσον αφορά θα πρέπει να εξετάσουμε τις εγκληματικές δραστηριότητε που έχουν διεθνές, διεθνή χαρακτήρα και δεν θα, θα πρέπει να εμποδίσουμε τη διάδοση παραποίηση των εμπορευμάτων, των φαρμάκων, των διαφόρων αγροτικών προϊόντων και τροφίμων στην Ευρωπαϊκή Ένωση καταπονηθεί. Τα ναρκωτικά είναι βασικό εισόδημα των κατομελών. Θα πρέπει να αντιμετωπιστεί μέσω μέτρων κατασταλτικών και προληπτικών. Μετά είναι τα συμφέροντα ε, εγκλημάτων ακόμα και γύρω από το στίχημα και ακόμα το γύρω από το νόμιμο στίχημα κερδίζουν οι εγκληματικές αυτές ομάδες. Θα πρέπει να υπάρξουν μέτρα πρόληψη και ε, καταπολέμησης. Η φορολογική παράδοση θα πρέπει να καταπολεμηθούν. Εκεί γίνεται ανακύκλωση του, του χρήματος που έχετε εγκληματικέ δραστηριότητε. Οπότε θα πρέπει να απαγορευτούν. Θα πρέπει να ρεύουμε τη συσχετισμό μεταξύ οργανωμένου κλίματος και τρομοκρατίας, σχέσεις που ίσως θα πρέπει να διερευνηθούν. Λοιπόν, μετά υπάρχει δίσδυση του οργανωμένου εγκλήματος, από ό,τι φαίνεται, στη διαχείριση των πόρων που διατίθεται στην, για την υποδοχή των μεταναστών. Φαινόματα διαφοράς και δίσδυση του οργανωμένου εγκλήματος και της μαφίας βρίσκεται επίσης διαχείριση των κέντρων υποδοχής ε, των ετούντων άσυλο. Έχει γίνει μια πραγματική business για αυτούς και επίσης και τα θέματα ανάθεσης υπεργολαβίας για τη δημιουργία αυτών των κέντρων υποδοχής ε, και επίσης των προσπαθειών για την ένταξη ε, των μεταναστών δημιουργούνται νέες δυνατότητες για την αγοράς για αυτούς τους εγκληματίες στην παροχή υπηρεσιών εκτός ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, για την υποδοχή των μεταναστών σε μια λύση. Λοιπόν, ε, επίσης εμπόριο ανθρώπων, εμπόριο οργάνων, πορνεία, δουλεία, το, έτσι χρησιμοποιούνται οι πρόσφυγες. Αυτή στιγμή χρησιμοποιούν εγκληματικές οργανώσεις. Άλλο θέμα. Είναι και η διαχείριση των αποβλήτων. Εκεί υπάρχει μεγάλος κίνδυνος να δυσδύσει το έγκλημα και είναι πολύ αποδοτική business για τους ε, εγκληματίες. Λοιπόν, τα τοξικά απόβλητα, η διαχείριση αυτών ε, επηρεάζει αρνητικά την νόμιμη αγορά και έχει καταστροφικά αποτελέσματα για τους πολίτες, ε, υπονομεύει το δικαίωμα της ζωής και της προστασίας της υγείας των πολιτών, η κακή διαχείριση των αποβλήτων και των τοξικών αποβλήτων. Χρειάζεται λοιπόν μία ε, έκθεση που προσπαθήσαμε να λάβουμε υπόψη τις διάφορες τροπολογίες. Ελπίζω να συνεχιστεί το πνεύμα συνεργασίας, ώστε να έχουμε ένα αποτέλεσμα τελικά που να μπορεί σημαντικά να συμμετάσχει ποιοτικά ε, στην αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος. Ε, ε, έχουμε χιλιάδες ομάδες οργανωμένου εγκλήματος κέντρα δύναμης ισχύω που επηρεάζουν τις νόμιες αγορές, τις πολιτικές και θεσμικές διεργασίες. Υπονομεύουν το κράτος δικαίου και τα θεμελιώδη δικαιώματα, αλλά μπορεί να επηρεάσει και την ποιότητα της ζωής, την οτροπία, τον πολιτισμό εκατομμυρίων Ευρωπαίων πολιτών ε, και διαφόρων κοινοτήτων. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θέλω να ευχαριστήσω και τους κοιόδους ηγητές, όλους εκείνους, όλους τους συναδέλφου που συμμετείχαν στις συζητήσεις. Ευχαριστώ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ευχαριστώ την Ευρωπόλ, την Eurojust το EPRS και όλους εκείνους που συνέβαλαν στην σύνταξη αυτής της έκθεσης. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε κυρία Φεράρα για την παρουσίαση της έκθεσής σας. Παρίστανται και κάποιοι σκιώδες ηγητές, προηγούνται στο χρόνο Ο κύριος Μέλο είναι ο σκιώδης ηγητής από το ΕΛΚΑ μέλο. Ευχαριστώ. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα κύριε Πρόεδρε να ευχαριστήσω την εισηγήτρια για την προσπάθεια που έκανε και την προσήλωσή της σε αυτό το θέμα. Η έκθεση πραγματικά έχει προτεραιότητα γιατί μας αγγίζει όλους και σίγουρα δικαιολογείται η προσπάθεια που θα καταβάλουν όλες οι πολιτικές ομάδες. Η διαφθορά είναι ένα περίπλοκο φαινόμενο, έχει κοινωνικές, πολιτικές, πολιτιστικές διαστάσεις σε όλες τις χώρες και γι' αυτό θα πρέπει ε, να λάβουμε υπόψη και τον διασυνοριακό χαρακτήρα που έχει και το οργανωμένο έγκλημα, τα σύνορα. Ε, ε, της εθνικής κυριαρχίας. Το άρθρο 83 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, απαιτεί κάποιους ελάχιστους κανόνες στα θέματα αυτά. Και στην συνήθι νομοθετική διαδικασία το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο μπορούν να θεσπίσουν ελάχιστους κανόνες για κάποια ποινικά εγκλήματα και κυρώσεις σε σοβαρό έγκλημα διασυνοριακού χαρακτήρα που προκύπτει από το χαρακτήρα ή τη συνέπειες αυτών των ε, παραβάσεων και την ανάγκη καταπολέμησής τους με κάποιες κοινέ βάσεις. Και αν αυτό που θεσπίζει ο νομοθέτης είναι ελάχιστοι κανόνες, θεωρώ ότι ε, οι πολίτες Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, περιμένουν από τους πολιτικούς ηθήνοντες μέγιστη προσήλωση παρά τους ελάχιστους κανόνες και μέγιστη δέσμευση στο στόχο αυτό. Γιατί μία από τι μάστιγες τη Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, είναι η διαφθορά. Υπάρχει διαφθορά και σε εθνικό και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Και η διαφθορά μερικέ φορέ αγγίζει και τα κοινοτικά κονδύλια. Και φτάνει σε μεγάλο βαθμό. Γιατί είναι πολύ ελκυστικό δόλο με αυτά τα κοινοτικά κονδύλια και χρειάζονται πολύ περισσότερε προσπάθειε για την πάταξη διαφθοράς από αυτές που έχουν γίνει μέχρι τώρα. Και φυσικά θέλω μια ανεξάρτητη Ευρωπαϊκή Εισαγγελική Αρχή με σαφώς καθορισμένες αρμοδιότητες και εξουσίες και ε, μια ενισχυμένη αστυνομική και δικαστική συνεργασία και πιο αποτελεσματική συνεργασία σε πανευρωπαϊκό επίπεδο επίσης είναι αποφασιστική σημασία και μάλιστα η στρατηγική για το 2020 στην εφαρμογή της και στην αποτελεσματικότητά της εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τον έλεγχο της διαφθοράς και να μην ξεχνούμε και το πολιτικό πλαίσιο που έχουμε αυτή τη στιγμή. Γνωρίζουμε ότι είχαμε μια χρηματοπιστωτική κρίση που αύξε την πίεση στις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις και θα ήταν να μην τι άλλο ένα αντιφατικό μήνυμα, να περιμένουν οι πολιτικοί στην Ευρωπαϊκή Ένωση από τις ε, κυβερνήσεις που ιδιαίτερα έχουν εφαρμόσει σκληρά μέτρα λιτότητας ε, να απαιτούν τέτοια μέτρα και η ίδια αυτή η πολιτική να είναι πιο χαλαρή στη χρησιμοποίηση των κοινοτικών κονδυλίων και δεν απαιτούν ε, παρόμοια αυστηρότητα στην εφαρμογή των πολιτικών πάταξης της διαφθοράς. Αντίστοιχη αυστηρότητα με αυτή στις πολιτικές λιτότητες. Η διαφθορά είναι υψηλή, προκαλεί τεράστιες ζημιέ, πολιτικέ, κοινωνικέ, οικονομικέ, ακόμη και περιβαλλοντικέ. Μα έδωσε το παράδειγμα η συγκεκριά. Και σα διαβεβαιώ ότι η ομάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματο θα σα στηρίξει και θα συνεργαστούμε μαζί σα ώστε να καταλήξουμε σε θετικέ και κατάλληλε λύσει. Σα διαβεβαιώ ότι θα είναι αμύωτο το ενδιαφέρον και η προσήλωσή μα προκειμένου να βρούμε μια ικανοποιητική λύση. Σας ευχαριστώ. Από τους σοσιαλιστές και δημοκράτες, η σκιώδη είναι η κυρία Γιώτοβα. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω την Λάουρα Φεράρα για την προσπάθειά της και τη συνεργασία που θα έχουμε. Να ευχαριστήσω και τους ε, συναδέλφους και οδησηγητές. Πιστεύω ότι είμαστε μια πολύ καλή ομάδα και θα φροντίσουμε όλοι να βρούμε κατάλληλες λύσεις. Έχουμε ήδη μια ιδέα για το τι σημαίνει διαφθορά σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Η έκθεση αυτή είναι πολύ σημαντική και με ενδιαφέρει ιδιαίτερος γιατί πριν από δύο χρόνια είχα ασχοληθεί με την έκθεση για Κουλίνο που είχε ένα παρόμοιο θέμα και γι' αυτό τα, ζητήματα αυτά με ενδιαφέρουν ιδιαίτερα. Με απογοήτευσε κάπως η στάση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην προηγούμενη έκθεση, γιατί περιμέναμε πολύ πιο ε, σημαντικές και αποτελεσματικές νομοθετικές προτάσεις ε, για την καταπολέμηση της διαφθοράς και του οργανωμένου εγκλήματος. Τώρα έχουμε μία διαφορά ως προς τους ορισμούς, γιατί αυτή τη στιγμή έχουμε ένα κοινό ορισμό για τη διαφθορά και η Λάουρα προτείνει και ένα κοινό ορισμό για το οργανωμένο έγκλημα. Χρειαζόμαστε τέτοιους ορισμούς κοινού, γιατί οι διαφορές μεταξύ των κρατών μελών οδηγούν και σε διαφορές στο ποινικό δίκαιο και σε διαφορετική αντιμετώπιση της καταπολέμησης της διαφθοράς και πολύ πιο δύσκολη λόγω των διαφορών. Περιμένουμε νομοθετικές προτάσεις και για την εναρμόνιση για τα θέματα της ε, σύγκρουσης συμφερόντων, τους φορολογικούς παραδείσους, ε, της, τη διοικητική διαφθορά. Δυστυχώς ε, μείναμε την όρεξη. Δεν έχει καταθέσει σχετικέ νομοθετικές προτάσεις ακόμη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Στην έκθεση για Κολίνο θέταμε μερικά πολύ εύστοχα ερωτήματα για το τι μέλη τι πρέπει να γίνει σε ευρωπαϊκό επίπεδο και ποια θα πρέπει να είναι η στάση των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων. Γιατί μέχρι στιγμή δεν έχουμε οριζόντια συνεργασία μεταξύ των κοινοτικών θεσμικών οργάνων. Το καθένα κάνει ό,τι θέλει. Θα πρέπει και μάλιστα το οργανωμένο έγκλημα εκμεταλλεύεται αυτή την έλλειψη συντονισμού και τα κενά. Το θέμα των δημοσίων συμβάσεων επίση είναι πολύ σημαντικό γιατί δημιουργεί ευκαιρίε για τους για, τη διαφθορά. Στη διαφθορά. Και έχουμε τέτοιες πρακτικές και ε, ακόμη και στο τομείο μετανάστευσης, ε, το τομείο για τους πρόσφυγες, τα κονδύλια που έχουν ε, προβλεφθεί για την προσφυγική κρίση. Το είδαμε και στην Κατάνια, όπου έγινε υπεξαίρεση κονδυλίων που προορίζονται για τους πρόσφυγες ε, με αποτέλεσμα το κανδύλι αυτά να καταλήξουν σε ιδιωτικές τσέπες. Ζητούσαμε λοιπόν νομοθετικές προτάσεις από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Μέχρι στιγμής που το μόνο που λάβαμε είναι μια έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη διαφθορά. Μια έκθεση που βρήθη πορισμάτων και συστάσεων, αλλά δεν υπάρχει καμία νομοθετική βάση για νομοθετική πρόταση. Περιμένουμε τη δεύτερη έκθεση τον Ιούνιο, αλλά δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη. Φαντάζομαι θα μας δώσει κάποιες εξηγήσεις για αυτές τις ολιγορίες η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Για να έχουμε έναν αποτελεσματικό αγώνα και πάταξη της διαφθοράς, χρειαζόμαστε παρόμοιους κανόνες στα κράτη-μέλη. Αλλά υπάρχουν διαφορετικοί τρόποι εποπτείας και ο μηχανισμός CVM για την Ρουμανία και Βουλγαρία δεν είναι πια αποτελεσματικός. Θεωρούμε ότι η καταπολέμηση της διαφθοράς μπορεί να γίνει πιο αποτελεσματική εφόσον γίνει εναρμονισμένα σε όλα τα κράτη-μέλη, χωρίς να στιγματίζουμε ή να στυλιτεύουμε την α ή τη β χώρα. Εμείς, σοσιαλιστές και δημοκράτες, θα καταθέσουμε συγκεκριμένες ε, τροπολογίες για την έκθεση. Είμαστε υπέρ της εναρμόνισης των νομοθετικών κανόνων και θα πρέπει να λάβουμε υπόψη και τη διαφθορά που γίνεται σχέση με τρίτες χώρες και όχι μόνο την ενδοκινοτική. Από τους συντηρητικούς και μεταρρυθμιστές, ο κύριος ε, Άντερσον. Να πω ότι ως ομάδα Υποστηρίζουμε την θέσπιση μια ευρωπαϊκή στρατηγική για την καταπολέμηση τη τρομοκρατία, του οργανωμένου εγκλήματο, του κυβέρνου εγκλήματο, του ξεπλήματο βρώμικου χρήματο. Άρα η αφετηρία μα είναι θετική. Και βλέπουμε στο σχέδιο έκθεση ότι Πράγματι προβλέπονται μια σειρά από σημαντικές πρωτοβουλίες όπως είναι η ενισχυμένη ανταλλαγή πληροφοριών, η καλύτερη συνεργασία στην επιβολή του νόμου μεταξύ των κρατών μιλιών, καλύτερη προστασία των ε, πληροφοριοδοτών, μεγαλύτερη διαφάνεια στη χρήση των ευρωπαϊκών κονδυλίων και ιδίω η σύνδεση μεταξύ οργανωμένου εγκλήματος, τρομοκρατίας και εμπορίας ανθρώπων για μας είναι πάρα πολύ σημαντικά ζητήματα, είναι θέματα που θα τα υποστηρίξουμε στην τελική έκθεση. Ωστόσο έχουμε κάποιες ανησυχίες, κάποιους προβληματισμούς ε, που είναι γνωστοί, όπως είναι η δημιουργία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, στην οποία εμείς αντιτιθέμεθα εξ αρχής και εμείς δεν υποστηρίζουμε η Ευρωπαϊκή Ένωση να γίνει μέλο της Γκρέκο και την, για την ανακατανομή των κονδυλίων ε, για κοινωνικούς σκοπούς. Για όλους αυτούς τους λόγους εμείς ε, ε, έχουμε αυτούς τους προβληματισμούς και θα προσέλθω στην διαπραγμάτευση που θα γίνει ε, με στόχο να τροποποιηθούν αυτά τα στοιχεία του σχεδίου έκθεσης ή και να αφαιρεθούν πλήρως, αλλά σε κάθε περίπτωση η στάση μου θα είναι υπηκοδοματική για να καταλήξουμε σε μια καλή έκθεση. Ευχαριστώ πολύ. Για τους φιλελευθέρους η Ναταλή Λοιπόν, καταρχάς θα ήθελα να ευχαριστήσω την κυρία Φεράρα για την ε, έκθεση αυτή που θεωρώ ότι είναι ιονή εξοχή διότι υπήρξε πάρα πολύ καλή συνεργασία και πολύ καλές συνεδριάσεις εργασίας μεταξύ Σκιωδών και Λάουρα Φεράρα. Πολύ, έλαβε πολύ καλά υπόψη σημαντικό ποσοστό των εκφραστέντων σχολείων που εμπλούτησαν το κείμενο. Ε, θα προσταθούν και κάποια άλλα κατά την περίοδο των τροπολογιών. Θα ήθελα να ευχαριστήσω διότι διοργάνωσε, χρησιμοποίησε ένα σημαντικότατο εργαλείο ενδιαφέροντα, ένα ερωτηματολόγιο ε, στα μέλη του Eurojust και τους διάφορους εισαγγελείς και στο συμβουλευτικό φόρουμ των ε, εισαγγελέων ε, και αυτό ήταν ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο που ήταν στη διάθεσή μας για να δημιουργήσουμε την έκθεση όσον αφορά το περιεχόμενο αυτό κάθε αυτό ε, τη μορφή του. Το σχέδιο εκθέσεως που προτείνεται ε, προτείνει αυτό λέμε προτείνει, εν πάση περιπτώσει το εφαρμόζουμε. Προτείνει λέγω μια προσέγγιση πρακτική. Δίνει προτεραιότητες. Αναφέρει στοιχεία. Μας συγκεντρώνει σε διάφορους τομείς. Για να μην έχουμε κάτι ανεξέλεγκτο με πάρα πολλές επιθυμίες που απομακρύνεται από το στόχο μας, επί της ουσίας. Υπογραμμίζουμε ότι πρέπει να εφαρμόζονται τα εργαλεία από τα κράτη-μέλη. Το επαναλαμβάνει αυτό η έκθεση. Θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι τα κάτι μελη ενσωματώνουν πολύ σωστά την ευρωπαϊκή νομοθεσία στην ένωμη τάξη τους και εφαρμόζουν τα εφιστάμενα ευρωπαϊκά εργαλεία και αν δεν γίνεται αυτό, να ξεκινά δικασίες κατά παράβαση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά αυτόν. Ένα στοιχείο άκρο θετικό στο σχέδιο εκθέσεως, με συγκεκριμένο, συγκεκριμένη στοχοθέτηση, είναι ότι υπογραμμίζει τη σχέση μεταξύ των φορολογικών παραδείσων και του ξεπλήματος βρώμικου χρήματος και την ανάγκη που υπάρχει εκεί να έχουμε ένα κείμενο που βελτιώνει την ανιχνευσιμότητα της ροής κεφαλαίων. Είναι κάτι πολύ επίκαιρο όπως γνωρίζουμε όλοι. Το υπενθύμησαν οι συνάδελφοι, πάντα το αναφέρουμε στις συζητήσεις μας εδώ στην Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών. Υπάρχει ανάγκη να δημιουργήσουμε Ευρωπαϊκή Εισαγγελία που δεν θα είναι μόνο ανεξάρτητη αλλά και ισχυρή. Ισχυρή και ανεξάρτητη. Ανεξάρτητη και ισχυρή. Μόνο έτσι θα προχωρήσουμε γρήγορα. Εν ονόματι της ομάδας μου θα ήθελα να επιμείνω επί τριών στοιχείων που θα μπορούσαν να εμπλουτίσουν το κείμενο πολέμηση κάθε μορφής εγκληματικότητας στον κυβερνοχώρο. Θα πρέπει να αναφέρεται ξεχωριστά ίσως τις κατηγορίες του, των προβλημάτων στους τομείς ειδικών παρεμβάσεων που αναφέρει το κείμενο. Διότι έχει βάρος η εγκληματικότητα στον κυβερνοχώρο, ε, παραποίηση προϊόντων, εξέπλημα χρήματος κλπ. Και είναι πολύ εντυπωσιακό το αποτέλεσμα. Είδα κάποια στοιχεία. 750 δισεκατομμύρια ευρώ στην Ευρώπη είναι το βάρος, το αποτέλεσμα αυτών των εγκληματικών δραστηριοτήτων. Έχουμε διασυνοριακό. 750 δισεκατομμύρια το χρόνο ευρώ μεγαλύτερο από το κόστος ε, κυκλοφορίας, αν θέλετε, ε, κοκαίνης, ηρωίνης και κάναβες. Μετά, έχει σημασία η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Θα πρέπει να έχει επαρκείς πόρους, ιδίους πόρους. Είναι πολύ σημαντικό για να πετυχάνει την αποστολή της και να έχει περισσότερες εξουσίες, να μην περιοριστικά την καταπολέμηση της ε, βλάβης των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τέλος, όσον αφορά την κατάσχεση το πάγωμα των ε, περιουσιακών στοιχείων, η οδηγία του ΙΧΑΣ 11 λειτουργεί, αρχίζει να δίδει καρπούς, αλλά τα σημερινά συμπεράσματα υπογραμμίζουν δύο στοιχεία που λείπουν. Τη δυνατότητα παγώματος και κατάσχεσης περιουσιακών στοιχείων ενός από τους συζύγους ή κληρονόμου σε περίπτωση καταδίκης δεν είναι αρκετά ακριβή σε διατύπωση. Στην πράξη βλέπουμε ότι όταν συμβαίνουν αυτά πολύ γρήγορα το χρήμα μεταφέρεται σε συγγενείς και έτσι εμποδίζεται κάθε δίωξη και είναι αδύνατον οι αστυνομικέ δυνάμεις και οι δικαστικές αρχές να κατάσχουν όλα αυτά τα βρώμικα χρήματα δεν μιλώ για κάτι αυτόματο, αλλά για δυνατότητα. Υπάρχει ένα είδος επικίνδυνης διαφυγής. Εγκληματικότητα και διαφθορά, οργανωμένο έγκλημα και διαφθορά, προφανώς κοστίζουν πάρα πολύ. Θα πρέπει λοιπόν να το προσμετρήσουμε και να εκμεταλλευτούμε αυτό το συσχετισμό για να δράσουμε, διότι πέραν αυτού όλα αυτά είναι μία απειλή για το κράτος δικαίου. Άρα θα πρέπει να βελτιώσουμε τη δυνατότητα πολιτικής απάντησης έναντι αυτών των πολυεθνικών εγκληματικών οργανώσεων που κινούνται σαν μπλοκάμια, απλών παντού τα μπλοκάμια τους. Αυτά και ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ε, και Ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, θέλω να συμφωνήσω με όσα είπε η Νάταλ Γκρίσμπεκ για τη συνεργασία των σκιωδών με τον εισηγητή σε διάφορες περιπτώσεις και τον ολοκληρωμένο τρόπο προετοιμασίας της έκθεσης. Ευχαριστώ την εισηγήτρια θερμότατα. Υπάρχουν διάφορα μηνύματα που συζητήσαμε στη διαδικασία ε, προετοιμασίας της έκθεσης. Να αποφύγουμε ε, μια μορφή χριστουγεννιάτικου δέντρου, για παράδειγμα, της έκθεσης, όπου θα αναδεικνύονται αυτά που ε, μας ενδιαφέρουν μεν, αλλά θα είναι τόσα πολλά που θα χάνονται. Από αυτή την άποψη η έκθεση πρέπει να είναι ευσύνοπτη. Ταυτόχρονα όμως θα πρέπει να αποφύγουμε την περίπτωση το Κοινοβούλιο να ε, κάνει κάποιες γενικές συστάσεις, να γίνει συζήτηση στην Ολομέλεια και το Συμβούλιο και η Κομισιόν να μας πούν ναι ευχαριστούμε πάρα πολύ και εμείς θα συνεχίσουμε τη δική μας δουλειά. Πρέπει να μπορέσουμε να καταλήξουμε σε συγκεκριμένα αποτελέσματα. Και από αυτή την άποψη εγώ θα υποβάλω αρκετές τροπολογίες για την έκθεση με κύριο στόχο να την καταστήσω πιο σαφή ως προς το ποιες είναι οι προσδοκίες μας από την Κομισιόν, το Συμβούλιο και τα κράτη-μέλη και μπορώ να σας δώσω και κάποια παραδείγματα. Για παράδειγμα, μιλάμε για την διαφθορά και βλέπουμε εδώ ότι η σύσταση που υπάρχει στην τρέχουσα, στο τρέχον σχέδιο έκθεσης έχει ξαναυπάρξει στο παρελθόν. Με ενοχλεί όμως το γεγονός ότι έχουν συσταθεί ε, focal points στα κράτη-μέλη. Έχουν γίνει σχετικές συζητήσεις στο Συμβούλιο και δεν βλέπω πουθενά κάποιο απτό αποτέλεσμα, ούτε κάποια πρόοδο να έχει σημειωθεί. Η Κομισιόν έχει μόνο μία φορά υποβάλει έκθεση για την καταπολέμηση διαφθοράς στα κράτη-μέλη και περιμένουμε τη δεύτερη. Και εγώ θέλω να είναι ολοκληρωμένη και θέλω να περιλαμβάνει και την καταπολέμηση διαφθοράς εντός των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων. Νομίζω λοιπόν από αυτή την άποψη ότι θα πρέπει να, τα αιτήματά μας να είναι πιο σαφή προς την Κομισιόν και στο Συμβούλιο και ότι δεν είμαστε διατεθειμένοι να κάνουμε γενικόλογες συζητήσεις και να καταρτίζουμε γενικόλογες συστάσεις προς την Κομισιόν. Θέλουμε συγκεκριμένα αποτελέσματα. Ο ΙΕ εξακολουθεί να ε, καταγγέλει την Ευρωπαϊκή Ένωση και συγκεκριμένα την Κομισιόν ότι δεν έχει ε, ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις που απορρέουν από την ε, Σύμβαση. Το ίδιο και με τον ε, ΟΣΑ, όπου διαπιστώνεται στην σχετική έκθεση ότι δεν υπάρχει επαρκής πολιτική βούληση για την καταπολέμηση της δωροδοκίας από επιχειρήσεις. Επίσης, πιστεύω ότι θα πρέπει να υπάρχει μια παράγραφος που θα αναφέρεται στο γεγονός ότι τα κράτη-μέλη δεν έχουν επαρκείς πόρους για να επιδιώξουν και να επιτύχουν τους στόχους που τίθενται. Υπάρχουν πάρα πολλές προτεραιότητες όπως είπαμε λοιπόν, αλλά θέλω η έκθεση αυτή να καταλήγει σε μια λίστα συγκεκριμένων προτάσεων για την Κομισιόν αλλά και για τα κράτη-μέλη, ώστε να μπορούμε να πούμε ότι διαφορά το τράφικιν, το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος ε, είναι οι τομείς που μα ενδιαφέρουν και διαπιστώνουμε ωστόσο ότι δεν έχει γίνει τίποτα. Πρέπει δηλαδή να πούμε ότι αφού θεσπίζουμε προτεραιότητες θα πρέπει να υπάρχουν και συγκεκριμένοι πόροι που θα, κατανέμονται για την προτεραιότητα αυτή και υπάρχει και ένας τομέας που έχει αγνοηθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχει οργανωμένο έγκλημα που εξειδικεύεται στην ε, ληστεία καταστημάτων. Χθε συναντήθηκα με τους εκπροσώπους των οργανώσεων των ε, λιανεμπόρων που μου είπαν ότι αυτό οδηγεί σε μεγάλες οικονομικές απώλειες για τους καταστηματάρχες και βεβαίως σε πολύ μεγάλα ψυχολογικά, ε, ψυχολογική, σε πολύ μεγάλη ψυχολογική πίεση για τους ε, υπαλλήλους. Η Europol έχει εντολή να συλλέγει τα σχετικά δεδομένα σε ε, εθνικό επίπεδο. Δεν δίνουν όμως προτεραιότητα σε αυτή τη διαδικασία. Και η ανάλυση που κάνει η Europol και το τι κάνουν οι εισαγγελείς δεν, δεν αξιοποιείται επαρκώς. Υπάρχουν, υπάρχει πολύ μεγάλη συλλογή πληροφοριών και δεδομένων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά αν ρωτήσει κανείς την Κομισιόν ε, πώς ε, έχουν συλλεχθεί όλες αυτές οι πληροφορίες και τα δεδομένα και πώς συνδέονται μεταξύ τους, ούτε καν η Κομισιόν δεν έχει ολοκληρωμένη εικόνα. Αυτά είναι σοβαρότατα προβλήματα που έχουμε σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν είναι το θέμα μόνο ε, ε, της, ε, της θέσης των προτεραιοτήτων. Ε, υπάρχει και πρόβλημα ως προς την επιδίωξη και ως προς την υλοποίηση των προτεραιοτήτων αυτών. Χρειαζόμαστε δεδομένα και χρειαζόμαστε να, να, να συλλέγουμε τα αναγκαία δεδομένα. Αυτά θα αφορούν ε, τις τροπολογίες μας ε, τις τροπολογίες που θα καταθέσω για το οργανωμένο έγκλημα, για το μεμονωμένο ε, έγκλημα, για την κατάσταση που επιδεινώνεται σε ορισμένες χώρες που θα μπορούσαν, για παράδειγμα, που θα μπορούσαν να αντιμετωπιστεί και με ε, αυστηρότερες ποινές. Επίσης υπάρχει ανάγκη να υπάρχει συνοχή στο ποινικό δίκαιο και να ε, διασυνδεθούν σε μεγαλύτερο βαθμό και οι διοικητικές διαδικασίες. Θεωρούμε ότι ε, οι κατηγορούμενοι έχουν ε, τα απαραίτητα ένδικα μέσα στα χέρια τους. Πώς εξασφαλίζεται η δίκαιη δίκη σε όλες τις περιπτώσεις. Αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικό θέμα για μένα, το γνωρίζει και η εισηγήτρια. Σε κάθε περίπτωση η στάση μου θα είναι επικοδομητική προκειμένου να βελτιώσουμε την έκθεση η οποία κατά την γνώμη μου είναι πάρα πολύ σημαντική. Ευχαριστώ πολύ. Χαίρομαι ιδιαίτερος για την ευκαιρία που έχουμε για εκτενή συζήτηση με συμμετοχή των σκιωτών εισηγητών και ευτυχώ έχουμε και την πολυτέλεια του χρόνου. Στις 12 πρέπει βέβαια να ξεκινήσουμε τις ψηφοφορίες Οπότε πρέπει να αρχίσουμε πια να προσέχουμε και το ρολόι. Αρκετοί συνάδελφοι ζήτησαν το λόγο. Τους παρακαλώ να είναι λακωνικοί. Γιάννα Άλμπρεχτ, είσαι και εκπρόσωπος ε, της ομάδας, γιατί άλλο όδη έχω για την ομάδα σου. Αν μπορείς να μας παρουσιάσεις και την άποψη των πρασίνων. Ευχαριστώ. Ναι, η Εύα Ζολή ε, κολλείεται σήμερα, γι' αυτό θα εκπροσωπήσω και τους πράσινους. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την κυρία Φεράρα για, το, ε, για την έκθεσή της μετά τις συστάσεις της Επιτροπής ΚΡΙΜ. Πολλές προσπάθειες πρέπει να γίνουν ακόμη για να καταπολεμήσουμε πιο αποτελεσματικά το οργανωμένο έγκλημα και όλες τις πτυχές της διαφθοράς. Ενδιαφέρουσα η δράση που προτείνει η συγκεντρία η θέσπιση ευρωπαϊκής νομοθεσίας για την καταπολέμηση περιβαλλοντικών εγκλημάτων, κατάργηση ή εξάλληψη των φορολογικών παραδείσων, γιατί ευνοούν το ξέπλυμα χρήματος και δέσμευση ή κατάσχεση των λογαριασμών και των περιουσιακών στοιχείων εγκληματικών οργανώσεων. Πριν από τρει εβδομάδε η ομάδα μα υπέβαλε μια πρόταση οδηγία για το θέμα αυτό και μετά το LuxLeaks και τα έγγραφα του Παναμά και τα συναφή σκάνδαλα Θεωρούμε ότι είναι κατεπίγον να λάβουμε κάποια δράση για τα θέματα αυτά. Ζητούμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή λοιπόν να υποβάλει το συντομότερο δυνατό μία πρόταση για τους φορολογικούς παραδείσους πέραν τη ε, εγκαθίδρυσης τη της Ευρωπαϊκής Αρχή, Αρχής που είναι αποτελεσματικό εργαλείο για την καταπολέμηση τη διαφθοράς και τη διασφάλισης των ε, κοινωτικών συμφερόντων θα πρέπει επιτέλου να ολοκληρώσουμε τι διαπραγματεύσει στο Συμβούλιο για να έχουμε μια πραγματικά ισχυρή και ανεξάρτητη Αγγελική Ευρωπαϊκή Αρχή για να μπορέσει μεταξύ άλλων να καταπολεμήσει και τη διαφθορά στο ΦΠΑ. Θα καταθέσουμε και σχετικέ τροπολογίε. Πάντω, χαιρετίζουμε το σχέδιο έκθεση γιατί αποτελεί μια στιβαρή βάση για τι περαιτέρω συζητήσει. Ευχαριστώ όλες και όλοι ήταν παρόντες ε, για τη συζήτηση. Κάτι που ενισχύει την αξιοπιστία της έκθεσης ε, και αποδεικνύει τη σπουδαιότητα της συζήτησης. Τρεις ε, ομιλητές έχουμε ακόμη και μετά θα ολοκληρώσω τον κατάλογο γιατί 12 πρέπει να περάσουμε στη ψηφοφορία. Σπινέλη, Σλάιν και Γκόμες είναι οι τρεις ομιλήτριες και ο κύριος Ράντεφ. Αλλά παρακαλώ θερμά να είστε επιγραμματικοί, γιατί πριν τις ψηφοφορίες έχουμε και ένα άλλο ζήτημα. Μπάρμπερα Σπινέλη, παρακαλώ. Ευχαριστώ την εισηγήτρια για την έξοχη παρουσίαση και διότι υπενθύμησε την δολοφονία του Τζοβάνι Φαλκόνε. Είναι, πολύ, είναι τόσο πιο σημαντικό να γνωριστεί η Ιταλική υπόθεση, να γίνει γνωστή η Ιταλική υπόθεση στην Ευρώπη στην προετοιμασία της εκθέσεως. Τι μας λέει λοιπόν η Ιταλική εμπειρία, ότι όταν η μαφία ε, στριμώχνεται, αισθάνεται άσχημα, σκοτώνει. Όταν τα πάει καλά, όπως σήμερα, σημαίνει ότι έχει δυσδύσει στις οικονομικές δραστηριότητες και στο δημόσιο τομέα. Και πιο συγκεκριμένα, στην Ιταλική πρωτεύουσα τη Ρώμη είναι σημαντικό να γνωρίζει ότι μία από τις ευρωπαϊκές ε, πρωτεύουσες είναι στα χέρια της μαφίας. Τώρα όσον αφορά κάποια, κάποιες τροπολογίες που θα ήθελα να υποβάλω συμπληρώντας την έξοχη παρουσίαση που έκανε η Λαόρα... Οι τοπολογίες αφορούν δύο σημεία. Πρώτα απ' όλα την εισαγγελία. Στην ομάδα μου δεν υπάρχει ένα ομόφωνο όραμα όσον αφορά τη εισαγγελία. Εγώ είμαι υπέρ μια ισχυρή ανεξάρτητης εισαγγελία. Υπενθυμίζω μόνο ότι υπάρχει μια τάση που έχει την πλειοψηφία στο Συμβούλιο να δημιουργηθεί ένας φορέας που θα συλλέγει με μαζικό τρόπο στοιχεία αδιακρίτως. Αυτό κατά την άποψή μου είναι ένας κίνδυνος προς αποφυγή. Διότι χωρίς ανάντι, ε, ε, συλλογή, ανάντι ε, διήθηση, συλλογή πληροφοριών κάτι κακό. Χαίρομαι όλος ιδιαίτερος που η Λάουρα ανέφερε το εξής. Αναφέρθηκε στον ορισμό της εγκληματικότητας στο δημόσιο και του εγκλήματος αντίσταση σε αυτή ε, στο ομαδικό έγκλημα. Υπάρχει λοιπόν και το αδίκημα συνδρομής ε, μιας εγκληματικής ομάδας ή ομάδας τύπου μαφίας. Αμφισβητείται πολύ το αδίκημα αυτό παρόλο που προβλέπεται από την νομοθεσία. Κατά την άποψή μου είναι σημαντική αυτή η έννοια να μπει στην έκθεσή μας και να συμπεριληφθεί στην Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Ε, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω πολύ θερμά τη συνάδελφο, την συγγήτρια, τη Λάουρα Φεράρα και όλους τους ε, σκιώδεις συγγητές για τη σημαντικότατη δουλειά που έκαναν. Πρώτα απ' όλα που υπενθύμησαν και όπως έκανε και η Βάρβαρα ε, τη δολοφονία του Τζοβάνι Φαλκόνη. Ε, να το υπενθυμίσουμε πρώτα απ' όλα σαν Ευρωπαίοι πριν το υπενθυμίσουν Ιταλοί. Και η Επιτροπή Κρίμα έκανε σημαντική δουλειά. Πρέπει να έχουμε επίγνωση τη σημασία τη ευρωπαϊκή διάσταση στην καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματο. Σήμερα οι μαφίε ε, αδιάφορα κερδοσκοπούν ει βάρο όλων των Ευρωπαίων. Εκμεταλλεύονται καλύτερα την ευρωπαϊκή ενιαία αγορά, καλύτερα από άλλου. Λοιπόν, ή θα, βρούμε, θα βρούμε στο ίδιο επίπεδο εργαλεία αποτελεσματικά να αντιταχθούμε σε αυτούς ή σε αυτό το παιχνίδι ήδη έχουμε χάσει. Πολύ καλή προσοχή που δίδεται στη καλύτερη εναρμόνιση την νομοθετική σε ευρωπαϊκό επίπεδο σε κοινό καθορισμό του οργανωμένου εγκλήματος και των σχετικών αδικημάτων και εγκλημάτων ε, ε, στα οικολογικά εγκλήματα, στα εγκλήματα που κινούνται μέσω της διαχείρισης των αποβλήτων κλπ. Θα πρέπει οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις να καταλάβουν ότι η δίστηση των μαφιών στην, στην νόμιμη οικονομία μας κάνει να χάνουμε απαραίτητους πόρους για να παρέχουμε και υπηρεσίες στους πολίτες μας. Ε, αυτό είναι ένα στοιχείο. Χρειάζεται καλύτερη δικαστική συνεργασία σε ευρωπαϊκό επίπεδο και όπως είπε ο Σάβος Κοράο, δυνάμεις αστυνομικέ έλεγαν ότι δεν μπορούν να συνεργαστούν αποτελεσματικά με τους Ευρωπαίους συναδέλφους για να αντιταχθούν σε ευρωπαϊκό επίπεδο στο φαινόμενο. Συμφωνώ όσον αφορά την ανάγκη να υπάρχει προστασία των πληροφοριοδοτών μέσω ευρωπαϊκής οδηγίας που καθορίζει σαφείς ελάχιστες προδιαγραφές, καταπολέμηση των φορολογικών παραδείσων που συνδέεται αυτό πολύ ε, στενά με το οργανωμένο έγκλημα και την ανακύκλωση χρημάτων. Χρειάζονται και εργαλεία παρακολούθησης και ελέγχου της χρήσης των ευρωπαϊκών πόρων και τη διαχείριση της υποδοχής των προσφύγων. Και το θέμα των τυχερών παιχνιδιών, εκεί θα έβαζα και κάτι άλλο, να προσέξουμε και το, το max fitting, δηλαδή το να στείνονται παιχνίδια, κάτι που κάνει πολύ η μαφία. Η κατάσχεση, κάτι που είπε και συνάδελφος των φιλελευθέρων. Η κατάσχεση είναι ένα εργαλείο πάρα πολύ σημαντικό. Περιμένουμε τη μελέτη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όσον αφορά τα ενδεχόμενα ωφέλη αν επεκτείνουμε το θέμα και στην κατάσχεση άνευ καταδίκης, όπως το βλέπει η Ιταλική νομοθεσία, ε, σεβόμενη τη δικονομία και τα δικαιώματα εκείνων που δικάζονται. Και θα πρέπει λοιπόν να ελπίζω και σε αυτό το τομέα να μπορέσουμε να προχωρήσουμε. Ευχαριστώ. Thank you very much, Σας ευχαριστώ, Έλλη. Η αναγκόμες τώρα. Ευχαριστώ. εκτιμώ ιδιαίτερω ε, που θα έχουμε την ευκαιρία να εκπονήσουμε τέτοια έκθεση και θα συμβάλλουμε και εμείς με τις τροπολογίε μας στο πολύ αξιόλογο έργο της κύρια Φεράρα. Πιστεύω, όπω και προλαλήσαντες, ότι σημαντικό θέμα είναι η νομοθεσία για τους του πληροφοριοδότες, στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελική Αρχή, τα εργαλεία για την κατάσχεση και δέσμευση περιουσιακών στοιχείων και τι θα έπρεπε τι θα πρέπει ήδη να κάνουμε για να κλείσουμε τα κενά και τα παραθυράκια και να καταπολεμήσουμε το ξέπλυμα χρήματος. Και νομίζω ότι δεν είναι μόνο θέμα της διείσδυσης της μαφίας από το οργανωμένο έγκλημα στην νόμιμη οικονομία. Είναι το πρόβλημα με τη διείσδυση της μαφίας στο πολιτικό μας κατεστημένο. Γιατί το οργανωμένο έγκλημα μερικέ φορέ κρατά σε ομοιρία τα κράτη μα Και οι μαφίε δεν ελέγχουν μόνο την οικονομία, ελέγχουν και το πολιτικό, την πολιτική εξουσία στα κράτη-μέλη, σε μερικά κράτη-μέλη, ε, σε πολλά κράτη-μέλη, σε πολλά θεσμικά όργανα, σε πολλά πολιτικά κόμματα. Και αυτό μας αποκάλυψε το σκάνδαλο με τα έγγραφα του Παναμά. Η φορολογική παράδειση δεν είναι μόνο παράδειση για φοροδιαφυγή και αποφυγή, φοροαποφυγή. Είναι παράδειση για την εγκληματικότητα και θα πρέπει να αντλήσουμε τα συμπεράσματα και τις συνέπειες αυτής της διαπίστωσης και να προστατεύσουμε όχι μόνο το τραπεζικό μας σύστημα ή να εμποδίσουμε τις τράπεζες αλλά και τον κλάδο που επιτρέπει στο τραπεζικό σύστημα να μετατραπεί σε μηχανισμό ξεπλήματος χρήματος. Νομίζω ότι αυτό είναι σημαντικό θέμα που πραγματεύεται η έκθεση και να αναπτύξουμε και διάφορα εργαλεία και κυρίως αυτό που θα θεσπίσουμε με τη Διερευνητική Επιτροπή που θα συστήσουμε για τη διαλεύκανση του σκανδάλου των εγγράφων του Παναμά. Πού είναι η έκθεση που μας υποσχέθηκε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη διαφθορά φέτος, πότε θα την καταθέσει επιτέλους. Δεν άκουσα και πολλά γι' αυτό. Περιμένουμε την έκθεση αυτή διακάως μετά την έκθεση του 2014 και ελπίζω να είναι πιο μεστή από την προηγούμενη και πιο εμπεριστατωμένη η νέα έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη Διαφθορά. Ευχαριστώ. Και τελευταίος ομιλητής μας, ο κύριος Ράντεφ. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε, έχουμε ναι. στην έκθεση επιτέλους κάποια μέτρα που τα ζητούσαμε εδώ και πολύ καιρό. Για παράδειγμα, ενίσχυση συνεργασίας ε, μεταξύ των αρχών επιβολής του νόμου, αστυνομίας και δικαστικού κλάδου, ενισχυμένους, ε, εναρμονισμένους κανόνες και μια ισχυρή και ανεξάρτητη Ευρωπαϊκή Εισαγγελική Αρχή είναι πολύ σημαντική για την ασφάλειά μας η καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος και της διαφθοράς. Είναι επίσης ε, σημαντικό αυτό το θέμα γιατί θέλουμε να βελτιώσουμε την καθημερινότητα των συμπολιτών μας και να νιώθουν ασφαλείς στις πόλεις ε, και στους τόπους που διαμένουν. Και αντίθετα θα πρέπει ανασφάλεια να νιώσουν οι εγκληματίε. Για να βελτιώσουμε λοιπόν την ασφάλεια των Ευρωπαίων πολιτών, εμείς εδώ στι Βρυξέλλες θα πρέπει να αρχίσουμε να εφαρμόσουμε μέτρα για να ενισχύσουμε την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Είμαστε εντό χρονοδιαγράμματος και θα ήθελα να ευχαριστήσω για άλλη μια φορά την Λάουρα Φεράρα για την εξαιρετική έκθεσή της. Ε, ε, έχει προετοιμαστεί πάρα πολύ καλά και Βεβαίως είναι σημαντικό το ότι αναφέρεται ο Τζοβάνι Βαλκόνη, αλλά όπως είπαν και οι σκιώδεις, θα πρέπει να επεκταθεί η έκθεση αυτή και να συμπεριλάβει τις προτεραιότητες της Επιτροπής μας και του Κοινοβουλίου για να μπορέσουμε να ε, καταλήξουμε σε μια συνεκτική έκθεση η οποία θα περιλαμβάνει πραγματικά σημαντικά στοιχεία. Ευχαριστώ όλους τους σκιώδες για τη συμβολή τους. Λάουρα, θέλεις να πεις κάτι πολύ σύντομα. Όχι. Οπότε, προθεσμή υποβολής τροπολογιών είναι 31 Μαΐου στις 12 το μεσημέρι. Ευχαριστώ όλους τους συναδέλφους που συμμετείχαν στη συζήτηση. Ένα ακόμη θέμα πριν περάσουμε στην ψηφοφορία στις 12 είναι η ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης προς την Επιτροπή της 29 η Ιανουαρίου από τον κύριο Κοράο για πιθανή παραβίαση των δικαιωμάτων των ασυνόδευτων αλλοδαπών αλληλίκων στη Σικελία. Σύμφωνα με τον κανονισμό μπορεί να υποβληθεί ερώτηση με έτοιμα γραπτής απάντησης προς την Κομισιόν και να συζητηθεί εδώ στην Επιτροπή σε περίπτωση που δεν έχει ε, ληφθεί απάντηση εντός της προθεσμίας. Ο κύριος Κοράου έστειλε την ερώτησή του στις 29 Ιανουαρίου του 2016 και σύμφωνα με, τον, με το άρθρο 130 Παράγραφος 5 του κανονισμού έπρεπε να είχε δοθεί απάντηση εντός 6 εβδομάδων. Η απάντηση αυτή δεν έχει ληφθεί, δεν έχει δοθεί απάντηση δηλαδή στο ερώτημα του κυρίου Κοράου. Οπότε κύριε Κοράου έχετε πολύ πολύ σύντομα το λόγο για να μας πείτε τι έχει συμβεί. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Στην Ιταλία και στην περιοχή μου στην περιοχή καταγωγή μου, στην Σικελία, έχουμε πολλού πρόσφυγες τελευταία χρόνια και είχαμε αύξηση τη παρουσίαση αλλοδαπών ανηλίκων ασυνόδευτων. Η Σικελία έχει περίπου 4.500 ανήλικα παιδιά. Προβλέπει τοπικό νόμο ότι ε, χρειάζεται να γίνει σωστή οργάνωση για τη στέγαση αυτών και να υπάρχουν και άτομα εκπαιδευμένα. 76 ευρώ το, ε, κοστίζει το κάθε παιδί, 45 είναι από το Υπουργείο Εσωτερικών και οι πληρώνουν τα υπόλοιπα. Δεν έχουν οι κοινότητε συγκελίε του πόρου για να καλύψουν το κόστος Οπότε ε, δεν μπορούν πλέον αυτοί οι χώροι φιλοξενίας να καλύψουν το κόστος για τα ανήλικα αυτά παιδιά. Είναι μια κατάσταση που δεν μπορούμε να τα διαχειριστούμε. Ε, λοιπόν, προτείνεται μια λύση για την περιοχή της Σικελίας. Να περάσουμε στα να μειώσουμε το κόστος από τα 76 στα 45 ευρώ. Ε, έτσι θα συμπιεστεί αναπόφευκτο το δικαίωμα των ανηλίκων. Αυτό που ζητούμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τέλος Ιανουαρίου είναι να λάβει επίγνωση του γεγονότος και είναι αποδεκτό ίσως ε, αν μπορούν να συμπιστούν τα δικαιώματα των ανηλίκων μειώνοντας τους σπόρους που διατίθενται σε αυτά, σε αυτά τα, στους χώρους φιλοξενίας των ανσυνοδεύτων ανηλίκων. Αυτό είναι το ερώτημα που έθεσα. Ευχαριστώ κύριε Κοράο, ευχαριστώ που υπήρξατε συνοπτικός. Ρώτησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, γνώριζε την κατάσταση και έθεσε και άλλες ερωτήσεις. Λοιπόν, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή που παρακαλώ να δώσει μια σύντομη απάντηση. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Καθυστερήσαμε αρκετά όσον αφορά την επεξεργασία του θέματος και τη γραπτής ερώτηση και λυπούμε θα απαργήσαμε να απαντήσουμε, θα προτιμούσαμε να μπορούσαμε σήμερα να ζητήσουμε συγγνώμη δίνοντας απαντήσεις στην ερώτηση που τέθη. Δυστυχώ η απάντηση ακόμα τελεί υπό επεξεργασία. Έχουμε επίγνωση ότι είναι πολύ λυπηρή αυτή η καθυστέρηση, διότι εκεί δημιουργείται μια κατάσταση πολύ σοβαρή. Κάνουμε τα πάντα τελικά το ταχύτερο να καταφτάσει η απάντηση και είμαστε διαθεσή σα για κάθε συμπληρωματική πληροφορία. Ευχαριστώ. Νομίζω ότι είναι λογική απάντηση την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Είναι πολύ σοβαρό το θέμα αυτό. Παραδεχτήκατε ότι υπάρχει καθυστέρηση και θα εξακολουθούμε να θέτουμε τα θέματα αυτά σοβαρών ερωτήσεων που καθυστερούν. Εντό ευλόγου χρονικού διαστήματο απαιτούνται απαιτήσει. Καταλαβαίνω ότι έχετε πιέσει. Υπήρχατε ειλικρινεί για το θέμα αυτό, για την ερώτηση αυτή. Και ε, θα πρέπει να δώσετε μια απάντηση στον κύριο Κοράου για πολύ σημαντικό ερώτημα για τους ασυνάδευτους ε, ανηλίκους. Φλέτα, ναι, πρώτο θέμα, λοιπόν, θα παρακολουθούμε το θέμα, θα δούμε πώς θα πάρουμε την... Ε, θα ενημερωθούμε και όταν λάβουμε την απάντηση. Θέλετε να προσθέσετε κάτι. Τι να, τι να προσθέσω, τι μπορώ να προσθέσω, Πρόεδρε. Ελπίζω να απαντήσουν σύντομα. Προσπαθούμε να βρούμε μηχανισμούς και έγκαιρα, διότι υπονομεύεται και αξιοπιστία των θεσμών αν δεν δίνουμε έγκαιρα ε, απαντήσεις. Ίσως στη διάσκεψη των Προέδρων ή σε σκόπιμο βήμα, σωστό βήμα, να βρούμε ένα μηχανισμό ώστε να λειτουργούν καλύτερα τα πράγματα και να έχουμε πιο βέβαιες ε, απαντήσεις και λύσεις. Όπως έτσι χρησιμοποιώ αυτό το μηχανισμό, περισσότερο από παλιά, για να υπάρχει σωστή, ο σωστός έλεγχος και η λογοδοσία. Σας ευχαριστώ και ευχαριστώ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την απάντηση. Περιμένουμε την απάντησή σας σε ευθέτω χρόνο. Καλό συνάδελφοι, μπορούμε να διακόψουμε για ένα τρίλεπτο ετοιμαζόμενοι για την ψηφοφορία που θα λάβει η χώρα στις 12. Ακριβώς. Α, τις κάρτες. Μην ξεχάσετε τις κάρτες. Φέρετε τις κάρτες αν δεν τις έχετε. colleagues, uh, please take your seats and we'll begin. Καθίστε παρακαλώ να ξεκινήσουμε την ψηφοφορία. Okay. So colleagues, uh, take your seats. Um, we begin the first... Ξεκινούμε με την πρώτη ψηφοφορία για τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια στη Θάλασσα, έγκριση του σχεδίου γνωμοδότησης. Μαζί με την πρόταση για σύνοροφυλακή και ακτοφυλακή, η Ευρωπαϊκή Κομισιόν υπέβαλε πρόταση για την τροποποίηση του οργανισμού που διέπει τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια στη Θάλασσα. Και σήμερα κάνουμε την ψηφοφορία για το θέμα αυτό. Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια στη Θάλασσα. Ψηφίζουμε για τη συμβαστική πρόταση. Ψηφίστε παρακαλώ. Has everyone voted? Ψήφισαν όλοι. Θα περιμένουμε λίγο μέχρι να ψηφίσουν όλοι οι συνάδελφοι. Και σημειώνουμε και την ψήφα του κ. Ντομάρα Διανατάσσω ισχυρό. τέλος 41. Όχι, συγγνώμη. Τελική ψηφοφορία. Ψηφίστε παρακαλώ. votes closed. Πέρας εγκρίνεται 44 υπέρ 7 κατά 0 αποχές συγχαρητήρια δεύτερη ψηφοφορία για το σχέδιο πρότασης για την Συμφωνία μεταξύ Ευρωπαϊκή Ένωση και Δημοκρατία του Περού σχετικά με την απαλλαγή από την υποχρέωση για τη διαμονή η ε, κυρία Γκάμπριελ. Ψηφίζουμε τη συμβαστική πρόταση. Ψηφίστε παρακαλώ. And the vote Τέλος Εγκρίνεται 50 υπέρ, 1 κατά, 1 κατά, 0 εποχέ. Δεν υπάρχει τελική ψηφοφορία. Αυτή ήταν. Και περι... περνάμε στην έκθεση σχετικά με την εφαρμογή τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ανθρώπων με αναπηρία, με ιδιαίτερη έμφαση στι καταληκτικέ παρατηρήσει τη Επιτροπή EPRD του ΟΗΕ. Μαρτίνα Άντερσον είναι η συντάκτρια τη γνωμοδότηση. Αν δεν έχετε αντίρρηση, περνάμε στην πληροφορία. Τροπολογία 2. Ψηφίστε παρακαλώ. Πέρας της εγκρίνεται. Τροπολογία 3. Ένας ψηφοφορίας. Πέρα στι ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 4. Ψηφίστε παρακαλώ. Πέρα στι ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 5. Ψηφίστε παρακαλώ. Πέρασε ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 6. Παρακαλώ. Πέρασε ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 7. Έναρξη της ψηφοφορίας. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 8 και 9. Ψηφίστε παρακαλώ. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Συμβαστική 8. Ψηφίστε παρακαλώ. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 11. Παρακαλώ ψηφίστε. Πέρας ψηφοφορίες. εγκρίνεται. Τροπολογία 12 ψηφίστε παρακαλώ. Πέρας ψηφοφορίες. εγκρίνεται. Τροπολογία 13 ψηφίζουμε. Πέρας ψηφοφορίες. εγκρίνεται. Τροπολογία 15 ψηφίστε παρακαλώ. Πέρας Εγκρίνεται. Τροπολογία 14. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 16. Ψηφίστε παρακαλώ. Πέρας. της ψηφοφορίες. Εγκρίνεται. Συμβεβαστική B. Ψηφίστε παρακαλώ. εγκρίνεται. Τροπολογία 20. Ψηφίστε παρακαλώ. Πέρας ψηφοφορίες. Εγκρίνεται. Τροπολογία 21. Έναρξη ψηφοφορίες. Τέλος της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 22. Ψηφίστε παρακαλώ. Πέρας ψηφοφορίας εγκρίνεται. Τροπολογία 23. Ψηφίστε παρακαλώ. Πέρας ψηφοφορίας εγκρίνεται. Ε, τροπολογία 24. Ένας ψηφοφορίας. Πέρας ψηφοφορίας εγκρίνεται. Τροπολογία 25. Ψηφίστε παρακαλώ. Πέρας εγκρίνεται. Τροπολογία 26, ένας ψηφοφορίας. Πέρας εγκρίνεται. 27, ψηφίζουμε. Πέρας ψηφοφορίας, εγκρίνεται. Συμβαστική πρόταση C. Ψηφίστε παρακαλώ. Πέρας εγκρίνεται. Ε, τροπολογία 35. Ένας ψηφοφορίας. Τέλος. Μάλλον όχι ακόμη. Τώρα τέλος. Εγκρίνεται. Συμβαστική δέλτα. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος. Εγκρίνεται. Ε, τροπολογία 38. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος. Υπάρχουν υπεράριθμοι στο ΕΛΚ. 2 τον αριθμό. Τέλος τώρα. Εγκρίνεται. Τροπολογία 39. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος, εγκρίνεται. Τροπολογία 40. άρχιτη ψηφοφορία. Τέλος, εγκρίνεται. 42. άρχιτη ψηφοφορία. Τέλος, εγκρίνεται. Συμβαστική ε, κατά τμήματα. Πρώτο τμήμα, άρχιτη ψηφοφορία. Τέλος. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα, άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος. Εγκρίνεται. Τροπολογία 43. Ή μάλλον 46. Πάμε κατευθείαν στη 46, άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος. Απορρίπτεται. Τροπολογία 47, άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος, εγκρίνεται. Τροπολογία 48, άρχεται η ψηφοφορία. Μήπως θέλετε να έχετε την 58, 48 με 58 να ψηφίσουμε από κοινού. Πολύ φαϊνή πρόταση. Ωραία προπολογίες 48 έως Σχεδόν θα Δεν ήταν και τόσο λαμπρή. Αλλά ας πέψουμε έστω και ξεχωριστά. 48 μόνο. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος. Εγκρίνεται. 49. Άρχεται η ψηφοφορία. τέλος εγκρίνεται 50 άρχεται ψηφοφορία τέλος εγκρίνεται 51 άρχεται ψηφοφορία τέλος εγκρίνεται 52 άρχεται ψηφοφορία τέλος Εγκρίνεται 53 άρχεται ψηφοφορία. Τέλος εγκρίνεται 54 άρχεται ψηφοφορία. Τέλος εγκρίνεται 55 άρχεται ψηφοφορία. <coughs> Τέλος. Εγκρίνεται. 56 άρχεται ψηφοφορία. Τέλος. Εγκρίνεται. 57 άρχεται ψηφοφορία. Τέλος. Εγκρίνεται. 58 άρχεται ψηφοφορία. Τέλος. Εγκρίνεται. 59 για διαγραφή. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος. 59 είπαμε. 59. Είστε κατά μάλιστα. Εγκρίνεται. 61. Άρχεται η ψηφοφορία. εγκρίνεται. 62 άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος εγκρίνεται. Αιτιολογικές σκέψεις. Τροπολογία 1 άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος εγκρίνεται και ψηφίζουμε το κείμενο όπως έχει τροποποιηθεί. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος, εγκρίνεται με 51 ψήφους υπέρ, μία κατά και δύο αποχές. Συγχαρητήρια στην εισηγητρία.